So, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann schlage ich vor, dass wir mit der Sitzung. και κύριοι, προτείνω να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην συνεδρίαση των συντονιστών αποφασίστηκε το ζήτημα της, ε, των σχολείων για την κυρία Γκερίνγκερ, για το trade sequences για την κυρία Γκαλό, για την ακόμη και την υπόθεση ασυλίας ο κύριος Ραπκάη, για τις γνωμοδοτήσεις συγκεκριμένα ζητήματα τεκμηρίου αθωότητας κυρία Τάιν, προσωρινή δικαστική συνδρομή Τσιόμπο, διαδικαστικές δικονομικές δικλείδες ασφαλείας για τα παιδιά έχει αναβληθεί. Τα λοιπά τρία θέματα έχουμε πει ότι δεν θα εκπονήσουμε γνωμοδότηση. Αυτό αποφάσισε η Επιτροπή, η, διά, Διάσκεψη των Συντονιστών. Για τα ε, οργανωμένα ταξίδια σε πακέτο, η αναβολή της ψηφοφορίας για να γίνει συζήτηση μεταξύ των ομάδων και άρα μεταφέρεται για τη 10η Φεβρουαρίου το θέμα αυτό. Αυτές ήταν ανακοινώσεις από τους συντονιστές. Και τώρα η έκθεση της κυρίας Γκέριγκερ Ντε κοινό σύστημα κοινό φορολογικό καθεστώς, το οποίο ισχύει για τις μετρικές και τις θηγατρικές εταιρείες διαφόρων κρατών μελών. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ε, Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η πρόταση του Συμβουλίου της 30 Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση του κοινού καταφορολογικού καθεστώτος για τις μητρικές και θηγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών καλύπτει ένα θέμα αρκετά περίπλοκο και σοβαρό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και γενικότερα. Προτείνονται λοιπόν διάφορα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος της φορολογικής βάσης, της εξουδετέρωσης λίγο πολύ της δυνατότητας φορολόγησης και της, εξουδε... της ε, φοροαποφυγής, δηλαδή την ε, διπλή φοροαποφυγή όπως τη λέμε, ε, διότι εμείς μπορεί να καταπολεμούμε τη φοροδιαφυγή, αλλά ε, μάλλον ε, μπορεί να καταπολεμούμε τη διπλή φορολόγηση μεταξύ κρατών μελών, αλλά υπάρχουν κάποιοι ξύπνοι οι οποίοι καταφέρνουν να αποφεύγουν σε διαφορετικές ένομες τάξεις να καταβάλουν το φόρο. Αυτό προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε την καταστρατήγηση δηλαδή της νομοθεσίας και την αξιοποίηση αποκλήσεων μεταξύ των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών, ώστε να μην επηρεάζεται αρνητικά η εσωτερική αγορά. Η διπλή φόρο αποφυγή λοιπόν πρέπει να αντιμετωπιστεί για να φέρουμε τα έσοδα ε, που χάνουν τα κράτη-μέλη και να αντιμετωπίσουμε τον αθέμητο φορολογικό ανταγωνισμό οι εκτιμούμενες ε, απώλειες από τους εθνικούς προπολογισμού είναι σημαντικές. Και κατά συνέπεια η φόρο αποφυγή ή η φορολογική παράδειση καλύπτονται σε έκθεση που έχει εκπονηθεί και αναφέρεται και στον δημοσιονομικό προγραμματισμό που υπολογίζει περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ με πολύ σημαντικές συνέπειες για την πενταετή περίοδο. Έτσι λοιπόν ε, θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε τις απώλειες από τα φορολογικά έσοδα σε πολύ ψηλά ποσά, δηλαδή ποσά τα οποία αντιστοιχούν βέβαια στους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Μετά τη θέση εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέτει μία έκθεση με αναφορά στην αποτελεσματικότητα της κατάργησης αυτών των, ε, παρα, των ε, ανισοτήτων στη φορολογία. Η δική μου η παρέμβαση έχει να κάνει με την διευκρίνηση της ε, διαδικασίας ώστε να καλυφθεί το θέμα της διπλής φόρου αποφυγής ή μη φορολόγησης. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς το λόγο, λέει ο Πρόεδρος. Όχι από ό,τι βλέπω. 27 Ιανουαρίου η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών στις 12 με ψηφοφορία στις 11 Φεβρουαρίου και ευχαριστώ κυρία Γκερίνγκερ Έτιγκερ. Και τώρα η κυρία Εύλην Ρέγνερ έχει παρακαλέσει το θέμα της να αναβληθεί. Μας μένει χρόνος περίπου 20 λεπτά και ρωτάω την γραμματεία τι μπορούμε ακόμα να κάνουμε. Έχουμε μόνο μια παρουσίαση για το πρωινό. πριν από τις προφορίες. Μας περισσεύουν 20 λεπτά. Καλώ, η γραμματεία μας λέει ότι δεν μπορεί να γίνει τώρα η παρουσίαση. Θα πρέπει να την αφήσουμε για το τέλος, μετά τις ε, ψηφοφορίες όπως έχει προγραμματιστεί. Ε, διακόπτουμε λοιπόν έως τις 10, όπου προβλέπονται οι ψηφοφορίες.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

Ja. Ja.

Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ,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

pourront Donc, euh, il y a six Oui, mais un truc alternatif, mais je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

So, ich denke, wir sind jetzt doch ziemlich... Νομίζω ότι είμαστε πλήρης τώρα. Έχουμε εκπροσώπηση για όλες τις ομάδες πλην μίας. Φαντάζομαι ότι θα καλυφθεί και αυτό. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν τις ψηφοφορίες και έχουμε πρώτα τις εκθέσεις του κυρίου Καρύμνα. με τριμέρη διάλογο που ολοκληρώθηκε. Ίσως θέλει να μας πει δύο λόγια κύριος Καρέμ. Πρώτα. Δεν έχουμε κατάλογο ψηφοφοριών. Κύριε Καρέμ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Can I um, start off first of all? Καταρχάς, να στείλω ένα μήνυμα ευχαριστίας, ευχαριστίων προς όλους που συνεργάστηκαν στην όλη διαδικασία. Σαφώς ήταν ε, περίπλοκο το ζήτημα για την Επιτροπή. Καταλήξαμε σε μία θέση που έχετε μπροστά σας για την ψηφοφορία. Ελάχιστα μέλη της Επιτροπής και ίσως και στο Κοινοβούλιο να μην γνωρίζουν κάποιες από τις προκλήσεις που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε για να φτάσουμε ως εδώ που φτάσαμε. Ελπίζω όμως ότι εδώ που φτάσαμε μπορούμε σήμερα να καταλήξουμε σε συμφωνία και ίσως αν όχι σήμερα στο Κοινοβούλιο να καταλήξουμε σε ισχυρή ε, πλειοψηφία που θα μας επιτρέψει να πετύχουμε τους στόχους μας. γενικόλογα αυτά που λέω, εκφράζομαι τι ούτω τρόπος, ούτως ώστε τα μέλη να καταλήξουν σε στήριξη του πακέτου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν θα κάνει άλλο το λόγο. Προχωρώ στην ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πρώτα, έχουμε του νόμου ελέγχου των ατήσεων λογαριασμών και ενοποιημένων λογαριασμών. Πρώτα έχουμε την οδηγία, μετά τον κανονισμό. Ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Έχετε όλοι τις κάρτες σας για την ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι 13 υπέρ, 8 κατά μία αποχή. Εγκρίνεται δεύτερη έκθεση του κυρίου Καρίμ και πάλι ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεκατρεις υπέρ, 8 κατά μία αποχή και εγκρίνεται συγχαρητήρια κύριε Καρίμ. Το επόμενό μας θέμα αφορά την έκθεση του αδέλφου Τσιέφκα. Θέλετε κάτι για να ξεκινήσουμε κύριε Τσιέφκα ή να πάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Καλώς. Τροπολογία 4. Δεν κάνουμε δηλώσει όπως πούμε, ξέρετε όλοι. Ψηφίζουμε το τεστ, τροπολογία 4 παρακαλώ υπέρ, κατά. εγκρίνεται 6 υπέρ κατά εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά εγκρίνεται. 1 υπέρ κατά εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά εγκρίνεται. 3 ε, υπέρ κατά εγκρίνεται το σύνολο για, με την ηλεκτρονική ψηφοφορία, το σύνολο της εκθέσεως. 22 υπέρ, χωρίς αποχές, χωρίς ψήφους κατά, εγκρίνεται. Ο νομισματικό νομοθετικό ψήφισμα, άρχεται ψηφοφορία. με 22 ψήφους χωρίς αποχέσεις και ψήφους κατά εγκρίνεται και τώρα η απόφαση για την χορήγηση της πραγματευτικής εντολής πάλι ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. πάλι με 22 ψήφους και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Καλή τύχη στις διαπραγματεύσεις. Το επόμενο θέμα είναι πάλι του κυρίου Καρίμ, επικουρικότητα και αναλογικότητα, 19η έκθεση σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας. Κύριε Καρίμ, θέλετε κάτι για να ξεκινήσουμε, αλλά η κυρία Γκερίνγκερ έχει κάτι να μας πει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα να επενθυμίσω κάτι σε όλους τους συναδέλφους ότι ο συμβιβασμός 3 δεν την χάνει υπό τη συμμετοχή τη ομάδας, της πολιτική ομάδα. Και γι' αυτό πιέζουμε να ψηφίσουμε. Την τροπολογία 40 και 41 δεν μπορεί να βασίζεται ο συμβιβασμός επί μιας τροπολογίας που δεν στηρίζεται από μια πολιτική ομάδα θα ήθελα κατά ξεχωριστά τμήματα να ψηφίσουμε την τροπολογία 40 και 41 διότι δεν, δεν αποτελούν τμήμα του συμβιβασμού. 41. Καλώς. Λοιπόν, έχουμε την πρόταση να ψηφιστούν τα 40 και 41. Υπάρχουν αντιρρήσεις από τον εισηγητή, όχι. Από ό,τι βλέπω, μπορούμε να ψηφίσουμε. Και προχωρώ. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 21 υπέρ κατά εγκρίνεται 1 υπέρ κατά εγκρίνεται 22 υπέρ κατά επαληθεύουμε ηλεκτρονικά την 22 8 υπέρ 14 κατά απορρίπτεται 23 υπέρ κατά εγκρίνεται υπαριθμόν ένα συμβαστική υπέρ κατά εγκρίνεται 19 της Επιτροπής Σταγματικών υπέρ κατά εγκρίνεται 25 υπέρ κατά απερίφθη 5 υπέρ κατά εγκρίνεται 6 υπέρ κατά εγκρίνεται 7 υπέρ κατά εγκρίνεται 20 υπέρ κατά εγκρίνεται 26 υπέρ κατά επαληθεύουμε 26 11 υπέρ, 11 κατά. Απερίφθη. 27 ταυτόσημη, 28 κατά. Απερίφθη. Καλύπτεται και 29, οι ε, παριθμόν 1 έω 18 τη Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων υπέρ, κατά. Επαληθεύουμε. 9 ε, ναι, υπέρ, 6 εποχές 7 ψήφοι κατά. 30 υπέρ, κατά. Απερίφθη, 8 υπέρ, κατά. Παλιθεύουμε. 8. Επαληθεύουμε. Έντεκα υπέρ, 11 κατά απερίφθη. Ε, συμβαστική 2 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, απερίφθη. 33 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 35 υπέρ, κατά, απερίφθη. 10 υπέρ, κατά, απερίφθη. 37 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η 38 έχει καλυφθεί. Συμβιβαστική. 4 από ό,τι λένε τα χαρτιά μου εδώ. Κάτι δεν πάει καλά. 3 έτσι. Στην 3 λοιπόν, συμβαστική 3 υπέρ. Κατά εγκρίνεται τώρα. Είπαμε θα ψηφίσουμε χωριστά 40 και 41. 40 πρώτα υπέρ, κατά. Απερίφθη 41 ταυτόσημη. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. 42 καλύπτονται, 43 υπέρ κατά, απερίφθη, 44 υπέρ, κατά εγκρίνεται, 45 και 46 υπέρ, κατά εγκρίνεται, 47 υπέρ, κατά απερίφθη, 48 υπέρ, κατά απερίφθη 49 υπέρ κατά εγκρίνεται συμβαστική 4 τώρα υπέρ κατά εγκρίνεται 51 υπέρ κατά εγκρίνεται 52-53 υπέρ κατά εγκρίνεται 54 υπέρ κατά εγκρίνεται 55 υπέρ κατά εγκρίνεται 56. Την έχουμε καλύψει νομίζω. 57 υπέρ κατά απερίφθη. 59 υπέρ κατά απερίφθη. 60 υπέρ κατά απερίφθη. 61 υπέρ κατά εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά απερίφθη. 63 υπέρ κατά απερίφθη. 64 υπέρ, κατά, απερίφθη, 66 υπέρ, κατά, απερίφθη, 67 υπέρ, κατά, απερίφθη, 68 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 13 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, συμβαστική 5 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 15 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 16 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 69 υπέρ, κατά, εγκρίνεται 17 υπέρ κατά απερίφθη 70 υπέρ κατά απερίφθη 71 υπέρ κατά απερίφθη 72 υπέρ κατά θαύμα 11 υπέρ, 11 κατά απερίφθη. 18 υπέρ, κατά εγκρίνεται 73 υπέρ κατά Απερίφθη. 19 υπέρ κατά εγκρίνεται 74 υπέρ κατά Απερίφθη. και τώρα το σύνολο της εκθέσεως ηλεκτρονικά παρακαλώ 14 υπέρ, 8 κατά, καμία αποχή και εγκρίνεται συγχαρητήρια κύριε Καρίμ. Και τώρα πάμε στην ετήσια έκθεση για τον έλεγχο τη εφαρμογή του δικαίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την κυρία Ρίχτεμπεργκερ. Ψηφίζουμε κατευθείαν. Ωραία. Τροπολογία υπάρχει μόνο ένα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. τρία, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Αύκο 3 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 5 26 υπέρ. Κατά. Περίφθη 27 υπέρ. 5 27 κατά. Επαληθεύουμε. 5 27. 10 υπέρ, 11 κατά, περίφθη. Αύκο 4 υπέρ κατά. Εγκρίνεται 5 12 υπέρ κατά. Απερίφθη 5 29 υπέρ κατά. Απερίφθη 13 5 υπέρ κατά. Απερίφθη 5 30 υπέρ κατά. Απερίφθη 5 31 υπέρ κατά. Επαληθεύουμε παρακαλώ 31 της πέτη 9 υπέρ, 12 κατά απερίφθη. Αύκο 2 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Αύκο 1 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 4 γκερίνγκερ υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 5 1 υπέρ. Κατά. Απερίφθη. 5 3 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 5 5 υπέρ. Κατά. Υπαλληθεύουμε. 9 υπέρ, 13 κατά, απερίφθη, 5 6 υπέρ, κατά, απερίφθη 7 υπέρ, κατά, απερίφθη 8 υπέρ, κατά, απερίφθη 5 9 υπέρ, κατά, απερίφθη 10 υπέρ, κατά, απερίφθη τροπολογία 5 υπέρ, κατά, εγκρίνεται τροπολογία 6 υπέρ, κατά, εγκρίνεται 7 κατά περίφθη 5-4 υπέρ κατά απερίφθη αύκο 5 υπέρ κατά επαληθεύουμε την αύκο 5 13 υπέρ, 9 κατά, εγκρίνεται, εύκο 6 υπέρ, κατά, απερίφθη, αύκο 7 υπέρ, κατά, απερίφθη, αύκο 8 υπέρ, Κατά. Επαληθεύουμε. Πέτη, ε, εγκρίνεται η ΑΦΚΟ 8. Εγκρίνεται. Ε, μπερδεύαμε κι εγώ. 5-17 παρακαλώ υπέρ κατά απεριφθεί 5-19 υπέρ κατά απερίφθη 28 πέτρι υπέρ κατά, απερίφθη 8 υπέρ κατά, εγκρίνεται 22 πέτυ υπέρ κατά, εγκρίνεται 5, 23 υπέρ κατά. Επαληθεύουμε την 23. Ε, Εννέα υπέρ 12 κατά περίπτωση. Πέτη 24 υπέρ κατά απερίφθη. 25 της πέτη υπέρ κατά απερίφθη. Πέτη 2 υπέρ κατά απερίφθη. 14 πέτη υπέρ κατά απερίφθη. 5,15 15 υπέρ κατά απερίφθη. 5,16 16 υπέρ κατά απερίφθη. 5,18 18 υπέρ κατά απερίφθη. Πέτη 11 υπέρ κατά απερίφθη. 5,20 20 υπέρ κατά επαληθεύουμε. Ναι, υπέρ, 13 κατά, απερίφθη 21 της 5 παρακαλώ, υπέρ, κατά, απερίφθη και ολοκληρώνουμε με την ονομαστική ψηφοφορία για το σύνολο του κειμένου ηλεκτρονικά. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια στην εισηγήτρια και περνώ στην έκθεση της κυρίας Καστέξ. Πείτε. Τέλει για αντίγραφα ιδιωτική χρήση. Πρώτα είναι η κυρία Καστέξ. Θα μα ε, μιλήσετε λίγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα θυμάστε ότι η έκθεση αυτή είχε αναβληθεί και δεν ψηφίστηκε στη Σύνοδο του Δεκεμβρίου και νομίζω ότι αυτό ήταν τελικά ωφέλιμο γιατί καταλήξαμε σε συμβαστικές τροπολογίες και ευχαριστώ την κυρία Νίμπλερ για την εξαιρετική συνεργασία μας από το Δεκέμβριο και νομίζω ότι τώρα καταλήγουμε σε μια ισορροπημένη έκθεση που θα αποτελέσει μια εξαιρετική συνεισφορά στις μελλοντικέ συζητήσει ε, για τη μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων του δημιουργού. Νομίζω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε λοιπόν. Θα ήθελα όμως ε, να προσθέσω ότι παρουσιάζω τρεις ε, τροπολογίες για το εκτιμώντας F βρίσκονται στο κατάλογο τροπολογιών, αλλά θα ήθελα να διαγράψουμε το 2010 για να το καταστήσουμε με την οδηγία 21. Κατόπιν έχουμε δύο προφορικές τροπολογίες, η μία για το εκτιμώντας Z και η άλλη για το άρθρο 6β σε σχέση με ένα πρόβλημα που δεν είχε αναφερθεί στην έκθεση και δεν υπήρχε καμία σχετική τροπολογία και μαζί με την ομάδα του ΕΛΚ προσέτουμε αυτή την αναφορά και κατόπιν έχουμε μία διαγραφή στο άρθρο 7α ε, λέει εκεί as far as the ultimate ε, consumer, the object being δηλαδή έχουμε τη διαγραφή αυτού του τμήματος της φράσης από το άρθρο 7. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Έξτρομ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να διαμαρτυρηθώ κατά αυτών των ε, λεγόμενων συμβαστικών τροπολογιών. Ε, το γραφείο μου τις έλαβε χτες στις 10 το βράδυ και πραγματικά δεν μπορούμε να εργαστούμε με τον τρόπο αυτό. Δεν ε, έχω τοποθετηθεί καθόλου για το θέμα αυτό. Έτσι λοιπόν αυτές είναι νέες τροπολογίες που έχει καταθέσει η κυρία Καστέξ μετά την τροπο... τη λήξη της προθεσμίας και δεν ακολουθούν τους κανόνες για συμβαστικές τροπολογίες εγώ ούτε καν ρωτήθηκα και μάλιστα βλέπω το όνομά μου στις τροπολογίες 2, 4 και 7 σε τρεις τροπολογίες ενώ δεν συμφωνώ με αυτές τις τροπολογίες γιατί ποτέ δεν με ρώτησαν, δεν μου ζήτησαν τη γνώμη μου και εδώ πραγματικά παραβιάζεται κάθε διαδικαστικός κανόνας για την τροπολογία 2, ε, τη συζητήσαμε το Δεκέμβριο και είχα πει σαφέστατα όχι και πάλι έχει κατατεθεί εδώ σαν να υποστηρίζει αυτό το συμβασμό. Έχω κάθετη αντίρρηση. Έτσι λοιπόν εγώ θα ήθελα αυτές τις αποκαλούμενες συμβαστικές τροπολογίες να τις θεωρήσουμε μη αποδεκτές γιατί έχουν κατατεθεί εκπρόθεσμα και ιδίω ε, τις τροπολογίες 2, 4 και 7 όπου βλέπω το όνομά μου κατά τη, παρά τη θέλησή μου. Και αυτές οι προφορικές τροπολογίες ήρθαν πάρα πολύ αργά, το ξαναλέω. Έτσι λοιπόν είμαι κατά όλων των προφορικών τροπολογιών ως θέμα αρχής, γιατί δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθούμε αυτή τη διαδικασία σε αυτή την Επιτροπή για την νομοθετούμε. Ευχαριστώ. Κυρία Βίξτρο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Υποστηρίζω όλα όσα είπε μόλις ο συνάδελφος και επίσης ε, και εγώ έχω συγχυστεί, αλλά ξέρετε, κάποιοι είναι πιο τυπικοί ε, και νομίζω ότι πρέπει να κάνω μία διευκρίνηση για την ψηφοφορία που θα κάνουμε για το φακέλο αυτό. Θέλω να υπογραμμίσω ότι οι μόνες ομάδες που έχουν κληθεί και συμμετάσχει σε αυτό το αποκαλούμενο συμβιβασμό είναι οι σοσιαλιστές και το ΕΛΚ και να πω ότι καμία από τις άλλες ομάδες δεν μπόρεσε να συμμετάσχει καν στις συζητήσεις. Ξέρετε, ποτέ κάτι τέτοιο δεν έχει ξαναγίνει σε αυτή την Επιτροπή και παρόλο που εμείς από τη δική μας πλευρά απευθυνθήκαμε στους σοσιαλιστές και δημοκράτες τουλάχιστον να έχουμε εμείς υπόλοιπη πρόσβαση στα συμβαστικά κείμενα αντί να συζητείτε αυτό αποκλειστικά μεταξύ συγγητρίας και της σκιώδους του ΕΛΚ. Δυστυχώς είχαμε συνεχή άρνηση από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Τελικά λάβαμε το κείμενο που θα συμφωνηθεί μεταξύ των δύο ομάδων χτες, γύρω στις 10 το βράδυ. Και ξέρετε τώρα, να βλέπουμε ότι τα ονόματά μας ε, είναι ε, μέρος ε, τροπολογιών, σαν έχουμε δεκτεί τροπολογίες τις οποίες το καν μας κάλεσαν να συμμετάσχουμε, δεν είναι σοβαρό. Και στο παρελθόν έχει φτάσει αργά ο καταλογός ε, της ψηφοφορίας και μάλιστα και για θέματα για τα οποία ήμουν υπεύθυνη εγώ. Αλλά εδώ βλέπουμε παντελή έλλειψη διαφάνειας. Είναι διαφορετικό λοιπόν το πρόβλημα γιατί σε άλλες περιπτώσεις συζητούσαμε μεταξύ μας όλοι οι συνάδελφοι, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν ακολουθήθηκε αυτή η διαδικασία. Από την αρχή είχαμε πει ότι δεν θα υποστηρίζαμε συμβαστικό κείμενο, καθώς οι θέσεις ε, της εισηγήτριας και των σκιωδών είναι αρκετά αποκλίνουσες, όμως καθώς τώρα φαίνεται ε, εδώ ε, ότι προτείνεται ε, σαν να υπάρχει ένα συμβιβασμό που συμφωνούν όλε οι ομάδε, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι ε, οι σοσιαλιστές εδώ έχουν ευθύνη και πολλές φορές έχουμε δει να γίνεται μια τέτοια διαδικασία, όμως εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικό όσοι ψηφίσουν να γνωρίζουν ότι κάποια μέλη δεν έχουν συμμετάσχει στις συζητήσεις για τους συμβιβασμούς και πραγματικά κάποιοι από εμά δεν έχουμε συμμετάσχει καθόλου και δεν υποστηρίζουμε κανένα από αυτούς τους συμβιβασμούς και νομίζω ότι αυτό ισχύει και για άλλες ομάδες πέρα από τη δική μας αλλά βέβαια δεν θα μιλήσω εξ τους. Λοιπόν, για να μην υπάρχει σύγχυση οι φιλελεύθεροι δεν έχουν καθόλου συμμετάσχει στην κατάρτιση αυτών των τροπολογιών, ούτε τις υποστηρίζουμε. Και επίσης αναμένω ότι για το μέλλον θα είμαστε ανοιχτοί και διαφανείς για το πώς γίνεται η διαδικασία και πώς εργαζόμαστε σε αυτή την Επιτροπή και σε αυτό τον Νίκο. Θα ήθελα να σας ζητήσω, Πρόεδρε, να θεωρήσετε απαράδεκτο ε, σε όλες αυτές τις αποκαλούμενες συμβαστικές τροπολογίες που καλύπτουν τα μέλη των φιλευθέρων 2, 3, 4, 7, 12 και 15. Κατά την άποψή μου είναι απαράδεκτες αυτές οι συμβαστικές τροπολογίες και έτσι θα πρέπει να δηλωθούν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Οι τροπολογίες, ε, εντάξει, φτάνουν καμιά φορά στις 10 το βράδυ. Έτσι έχουν τα πράγματα, το δεχόμαστε. Όμως, άλλα θέματα που τέθηκαν από τους δύο συναδέλφους ε, θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρά. Και μπορώ να σας πω, από τη σκοπιά της δικής μου ομάδας, εμείς δεν έχουμε συμμετάσχει σε καμία διαπραγμάτευση από αυτές που έλαβαν χώρα για αυτές τις ε, συμβαστικές τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Στη βάση αυτή υποχρεούμε να υποστηρίξω και τους δύο συναδέλφους που πήραν το λόγο τελευταία. Ευχαριστώ. Κύριε Σπερώνη, ευχαριστώ. Και εγώ υποστηρίζω τους συναδέλφους που πήραν το λόγο πιο πριν. Ε, θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση σύμφωνα και με το όσο είπε ο κύριος Κάρεμεν. Ναι, είναι πράγματα που συμβαίνουν αυτά στη ζωή. Δεν μπορεί κάποιος να αποφύγει μία ασθένεια, παραδείγματο χάρη. Όμως ε, το να κατατίθεται τροπολογία στις 10 το βράδυ είναι κάτι που δεν γίνεται. Κύριε Καστέξ, παρακαλώ. Ε, πραγματικά με εκπλήσουν οι παρεμβάσεις των συναδέλφων να υπενθυμίσω ότι πραγματοποιήσαμε πολλές συνεδριάσεις με τους σκιώδεις εισηγητές και όλοι οι σκιώδεις εισηγητές είχαν ε, κληθεί και η ομάδα των πράσινων και η ομάδα των φιλελευθέρων στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις. Και εγώ ενώ είχα προτείνει να εργαστούμε ε, επί διάφορων σημείων και να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε, συνολικά αυτοί απέρριψαν την πρόταση και είχαν αντιτεθεί στο σύνολο της έκθεσης σε τέτοιο βαθμό που δεν υπήρχε δυνατότητα να καταλήξουμε σε κοινούς συμβιβασμούς. Παρόλα αυτά, Καθ' όλη την περίοδο πριν από την ψηφορία που είχε προβλεφθεί το Δεκέμβριο είχαν ενημερωθεί για τις συμβαστικές τροπολογίες. Είχατε λάβει αυτές τις τροπολογίες και είναι και μάρτυρα σε γραμματεία. Είχατε λάβει αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες τις οποίες είχατε συμμετάσχει και δεν είχατε ενημερώσει ότι δεν λάβατε τις τροπολογίες. Έτσι λοιπόν συνεχίσαμε το έργο μας με τις ομάδες που συμφωνούσαν για την αναζήτηση τροπολογιών για τα θέματα αυτά. Οι συμβαστικές τροπολογίες έφτασαν χτες το βράδυ ε, στις 5 το απόγευμα. Είναι αλήθεια ότι καθυστέρησε λίγο περισσότερο ο κατάλογος των ψηφοριών γιατί καταλήξαμε συμβασμό στις 5 το απόγευμα. Τώρα, σε σχέση με τα διάφορα στοιχεία, εγώ διαφωνώ μαζί σας και πιστεύω ότι υπήρχαν κάποιε από τι τροπολογίε σα που ήταν θετικέ. Και στον κατάλογο των ψηφοριών υπάρχουν κάποιε από τι τροπολογίε σα όπου έχω βάλει συν. Εδώ τώρα μου αμφισβητείτε το δικαίωμα να μπλουτίσω την έκθεσή μου με ορισμένα από τα στοιχεία που είχατε καταθέσει εσείς στις δικές σας τροπολογίες. Δεν ε, βλέπω να είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Εγώ έκανα μία πρόταση ε, όπου αναφέρεστε. Μπορείτε πολύ καλά να καταψηφίσετε αυτή την συμβιβαστική πρόταση. Μπορείτε να ζητήσετε να ψηφιστούν ξεχωριστά οι δικές σας τροπολογίες, αλλά δεν μπορείτε να μου αρνηθείτε το δικαίωμα ε, να υπερψηφίσω για την τροπολογία 5, παραδείγματο χάρη, ακόμη και αν υπάρχει το όνομά σα επάνω, είναι μια λογική διαδικασία. Εγώ έλαβα υπόψη όλε τι συνεισφορέ, ακόμη και αν είστε αντίθετοι στην έκθεσή μου στο σύνολό τη. Ευχαριστώ. Η κυρία Νίμπλερ, η κυρία Έγκστρομ και μετά μπορούμε να αποφασίσουμε. Η κυρία Νίμπλερ, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρακολουθώ τη συζήτηση. Δεν θέλω να τοποθετηθώ επί τη διαδικασία γιατί δεν ξέρω πώς ε, ε, προχώρησε η ψηφοφορία, ο προσδιορισμό των θέσεων με την κυρία Καστέτσικα και τις άλλες ε, ομάδε, αλλά θα προτείνω εφόσον τρει από τι ομάδε μα λένε ότι δεν είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να δούνε καν τις συμβαστικές τροπολογίες, τροπολογίες θα έλεγα να αναβάλουμε την ψηφοφορία δεν έχει κανένα νόημα. Και δεν δίνει και καθόλου καλή εικόνα το να φαίνεται ότι οι δύο μεγάλες ομάδες ρύθμισαν το θέμα αυτό μεταξύ τους με τις μυριστικές τροπολογίες. Θα ήταν μια κίνηση καλή θέληση εναντί των μικρότερων ομάδων. Έχουμε καθυστερήσει ήδη. Εγώ προτιμούσα στις 17 Δεκεμβρίου να γίνει ψηφοφορία, αλλά δεν είχαμε συμβαστικές ψηφοφορίες. Τώρα λοιπόν Γι' αυτό προτείνω πριν ε, αρχίσουμε να συζητάμε καλύπτεται δεν καλύπτεται ε, και χάσουμε χρόνο με αυτό και ταλαιπωρηθούμε να, να αναβάλουμε για να γίνει πιο σωστά η δουλειά. Επισήμως λοιπόν κατά αυτό το αίτημα για αναβολή της ψηφοφορίας. Έγκστρομ και μετά Καστέξ. Βέβαια, είστε πρόσδεκτοι να υπερψηφίσετε οδήποτε τροπολογία μου. Εγώ θα συνέστηνα να υπερψηφίσετε όλες. That is not the Δεν έγκυται εδώ το πρόβλημα. Το πρόβλημά μου είναι ότι μου δίνετε πράγματα, μου παρουσιάσετε πράγματα ως συμβιβασμούς με την υποστήριξή μου όταν δεν μου μιλήσατε καν. Και σίγουρα δεν έχετε την υποστήριξή μου. Αυτό με προβληματίζει, σε αυτό προβάλλω αντίρρηση και γι' αυτό όλες οι βαστικές αστροπολογίες δεν θα πρέπει να είναι παραδεκτές. Καλώς. Έχουμε όμως ούτως ή άλλως ένα έτοιμα για αναβολή. Να σας εξηγήσω και εγώ τις δικές μου θέσεις. Έχουμε. Κυρία Καστέξ, θέλετε πρώτα να μιλήσετε εσείς. Καλά. Κοιτάξτε, λοιπόν, είμαι αντίθετη στην αναβολή της εκθέσεως, της ψηφοφορίας. Επανειλημμένα είχε αναβληθεί με η συζήτηση της στην ημερήσια διάταξη και το Δεκέμβριο είχα μια αναβολή, πετύχα μια ισορροπία δεν νομίζω ότι πρέπει να δημιουργείται προηγούμενο δεν είναι προηγούμενο να γίνω την παραμονή ο φοριών κλπ. Έχω εμπειρία εδώ για να ξέρω ότι αυτό πολύ συχνά συμβαίνει, δεν είναι κάτι ασύνηθες και είμαι αντίθετος σε αυτό που λέει ο κύριος Έγκστρομ. Συμμετείχαν σε δύο συνεδριάσεις τεχνικής ε, φύσεως των σκιωδών και ε, συνεργαστήκαμε για συμβιβασμούς τόσον αφορά τις συμβαστικές τροπολογίες που συμπεριλαμβάνουν στοιχεία των τροπολογιών τους νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάναμε αυτό που έλεγε η Λίδια ψηφίζουμε συμβαστική τροπολογία είναι δική μου ευθύνη να παρουσιάσω συμβαστικές τροπολογίες και αν απορριφθεί μπορούμε να ψηφίσουμε ξεχωριστά τις τροπολογίες ε, που έχουν συμπεριληφθεί Αυτά προτείνω διαδικαστικά να κάνουμε. Καλώ. Όλοι υπάρχει το αίτημα για την αναβολή. Πρέπει να αποφασίσουμε. Θα θέλω όμως να μιλήσω για το παραδεκτό πρώτα. Γιατί κοιτάξαμε το άρθρο 161.4 του κανονισμού που έχει με πλάγιες γραμμές ένα κείμενο, μία παράγραφο, αυτό δείχνει ότι έχει απασχολήσει την Επιτροπή των Σταματικών Υποθέσεων, όπου γίνεται λόγος για τις συμβαστικές τροπολογίες, για το πώς θα ληφθεί η απόφαση και για το ποιος καταθέτει τις συμβαστικές τροπολογίες. Αναφέρεται λοιπόν ότι συμβαστικές τροπολογίες καταθέτουν οι ομάδες, δεν λέει όλες οι ομάδες, άρα θα μπορούσε ακόμη και η μειονότητα των ομάδων να καταθέσει τις συμβαστικές τροπολογίες. Εάν πρόκειται όμως να κατατεθεί ως προς την ερμηνεία της ΑΦΚΟ μια ένσταση για την κάθε από, μία από τις συμβαστικές τροπολογίες, θα έπρεπε αυτό να το ψηφίζουμε σε κάθε περίπτωση. Έχουμε αίτηση λοιπόν για αναβολή της ψηφοφορίας από την κυρία Νίμπλερ. Εάν την εγκρίνεται με την ψηφοφορία θα ψηφίσουμε την επόμενη συνεδρίαση. Εάν δεν την εγκρίνεται τότε θα πρέπει να προβάλλεται ένσταση σε κάθε περίπτωση συμβαστική και αναλόγως να γίνεται ψηφοφορία για την έγκριση της ένστασης σημεί. Τώρα ψηφίζω την ψηφοφορία για την αναβολή, την πρόταση κυρίας Νίμπλερ. Ποιος είναι υπέρ της αναβολής της ψηφοφορίας. Κατά Εγκρίνεται λοιπόν η αναβολή για την προσεχή συνεδρίαση της ψηφοφορίας. Και έτσι η έκθεση κυρίας Καστέξ, παρακαλώ έχετε το λόγο. Κοιτάξτε, είναι άχρηστη αυτή η αναβολή, αυτό πιστεύω. Και διαπιστώνω ότι πραγματικά υπάρχει βούληση σαμποτάζ κατά της εκθέσεως αυτής. Ωστόσο, Σα επισημαίνω ότι αποφασίστηκε στην προσοχή συναντήση να ψηφίσουμε, λέει ο πρόεδρος. Και τώρα έχω την έκθεση του κυρίου Ραπκάι. 50. Επιτροπή Οικονομικών, έχετε το λόγο. Κύριος Ραπκάι, μια και έγινε συζήτηση όπως έγινε μόλις τώρα, έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις, ξεκινώντας, πριν περάσουμε στην ψηφοφορία για τη δική μου έκθεση. Η πρώτη παρατήρηση είναι εξή. Και ξεκινώ ως εξή. Θυμάμαι με χαρά μια συζήτηση πριν από δύο ώρες ή λιγότερο ακόμα μεταξύ των συντονιστών όπου είπαμε ότι σε γνωμοδοτήσεις ε, θα πρέπει να, θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε στις δικές μας αρμοδιότητες ως Επιτροπής. Και θα θυμάστε ότι ακριβώς αυτό πρότεινα και ως εκ τούτου προσάρμοσα και την πρόταση εκθεσεώς μου σε αυτό το στόχο. Ακριβώς δηλαδή στους τομείς ο οποίος έχει αρμοδιότητα επί της ουσίας η δική μας Επιτροπή. Από την άλλη, κάθε συνάδελφος, κάθε ένας και κάθε μία από εμά μπορεί να τοποθετηθεί με τις τροπολογίες του σε ό,τι βούλεται, όπως συνέβη και επειδή ακούστηκαν κάποια ψιθυρίσματα με επικρίσεις για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκα την έκθεση, εδώ συνέπεια της επιλογής μου αυτής, να περιοριστώ δηλαδή στην κατουσία αρμοδιότητα της Επιτροπής μου, είναι και ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκα τις συμβαστικές τροπολογίες. Δηλαδή πάλι τις ε, συμπυκνώνω έτσι ώστε να αναφέρονται μόνο σε ζητήματα καθήλυνα αρμοδιότητας της Επιτροπής των Νομικών Υποθέσεων. Δεν έχει νόημα να επεκταθούμε και να πλατιάζουμε και να μιλάμε για πράγματα για τα οποία ούτως ή άλλως έχει ήδη εγκρίνει η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή ή τα απορρίπτει. Λοιπόν, ας μην πάμε εκεί που δεν έχουμε αρμοδιότητες, ας μην πάμε εκεί που ξεπερνούμε τις αρμοδιότητές μας και παρακαλώ θα το πω και ξεκάθαρα για κάθε άλλη επιτροπή, καλό είναι να κάνει το ίδιο γιατί ε, είναι όρος και προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα των εργασιών του Κοινοβουλίου η κάθε καθήλυνα αρμόδια επιτροπή να κάνει τη δουλειά της στον τομέα των αρμοδιοτήτων της και να μην μπαίνουν στα χωράφια της όλες οι άλλες, γιατί θα είναι εκατοντάδες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες θα είναι συναρμόδιες κάποιες επιτροπές για γνωμοδότηση και δεν θα πρέπει να μπαίνουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της κύριας επιτροπής. Αυτό λοιπόν, να επικεντρωθούμε στη δουλειά μας. Πρώτον. Δεύτερον, και είναι και σχετικό βέβαια, η έκθεσή μου, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ή τουλάχιστον άκουσα από χθε με τις διαπραγματεύσεις ε, και σήμερα το πρωί ακόμη, δεν έχει μεριμνήσει η επαρκώς δεν έχει ληφθεί απαραίτητη μέρημνα για την αποστολή των καταλόγων των ψηφοφοριών. Και αυτό δεν αφορά το δικό μου γραφείο, γιατί δεν το στέλνει το δικό μου γραφείο, ε, δεν στέλνει τους καταλόγους των ψηφοφοριών το δικό μου γραφείο, αλλά αντελήφθην ότι τελευταία στιγμή και υποποίηση χρειάστηκε να εργαστεί η ε, γραμματεία της Επιτροπής εχθές ε, αν λοιπόν μπορέσουμε να κάνουμε πιο οργανωμένα και συντονισμένα τη δουλειά μα, ίσω να, να μην αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα στο μέλλον. Σημειώνω λοιπόν ότι δεν οφείλεται στο δικό μου γραφείο αυτή η εσπευσμένη αποστολή των ε, καταλόγων ψηφοφοριών. Δεν θέλω να καταδικάσω κανέναν ούτε να επικρίνω κανέναν. Ξέρω ότι είναι δύσκολη η δουλειά αυτή και ότι είναι ε, περίπλοκο όταν έχουμε τόσο μακροσκελείς καταλόγους ψηφοφοριών και θέματα μεγάλα και διεξοδικά να είμαστε και στο χρόνο ε, στην ώρα μας έτοιμοι. Ο κύριος Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Έκανε φυή εργασία και ανοιχτή ο εισηγητής και συμβάλαμε κατά σημαντικό τρόπο για να καταλήξουμε σε μια ισορροπημένη απόφαση. Όμως Παίρνω το λόγο και δράτω με τις ευκαιρίες για να εκφράσω μία θέση μου που έχω εκφράσει και προηγουμένως. Άρθρο 7 και άρθρο 11. Είναι δύο ζητήματα που δεν είναι μόνο ειδική αρμοδιότητα, όπως ξέρει ο, ο εισηγητής της Νομικής Επιτροπής, αλλά της Οικονομικής. Όμως αυτή τη ψηφοφορία τη βλέπω με προβληματισμό, κυρίως όσον αφορά τροπολογία 96 για το άρθρο 7 και τροπολογία 115 που αφορά το άρθρο 11 Θεωρώ λοιπόν ότι μπορεί να αποτελεί και ένα είδος μήνυμα προς την Οικονομική Επιτροπή. Η διαγραφή του άρθρου 7 θα αλλάξει την ισορροπία μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και της ισορροπίας, γιατί θα επέτρεπε ε, την, ε, τη, αλλάζει τη φιλοσοφία της ε, νομοθεσίας για το βάρος απόδειξης. Δηλαδή η αρχή, η ελεγκτική αποδυναμώνεται ε, και δεν προστατεύονται παρκώς τα θύματα. Όσον αφορά το άρθρο 11, πιστεύω ότι τα θύματα... Ξέρουμε ότι υπάρχει το δικαίωμα του ανταγωνισμού, έτσι. Ίσως να υπάρχει κάποια συμμετρία όσον αφορά την ενημέρωση. Κάποιος που είναι θύμα παραβίασης του νόμου δεν γνωρίζει ότι είναι θύμα πριν να είναι θύμα. Μέσω των προγραμμάτων που ευνοούν τις επιχειρήσεις Επιτρέπεται λοιπόν στα θύματα να γνωρίζουν ότι υπάρχει ε, καρτέλα από επιχειρήσεις και να, ε, μάλλον να μπορεί να ζητήσουν αποζημίωση. Και τα εθνικά δικαστήρια μπορούν να αποφασίσουν το είδος αποζημίωσης για τις μεταδόσεις που πρέπει να πληρωθούν. Έχουν δυνατότητα οι δικαστές να κάνουν επαλήθευση. Αν μπορούν να πληρώσουν αυτοί που διέπραξαν την παράβαση και ποιο ποσό οφείλεται σε κάθε επιχείρηση. Αν διαγραφεί παραγράφους, θα υπονομευθεί η σωστή λειτουργία του μηχανισμού. Εκφράζω επιφυλάξεις επί των σημείων αυτών, διότι όσον αφορά το σύνολο του κειμένου νομίζω ότι έχουμε πετύχει μια σωστή ισορροπία. Κάθλο, σημειώνουμε τις επιφυλάξεις, όμως πρέπει να ψηφίσουμε τώρα και τώρα πάω στην τροπολογία 20, 50 ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 51 υπέρ, κατά. Επαληθεύουμε την 51 παρακαλώ υπέρ, άρχιτη ψηφοφορία. 12 υπέρ, 9 κατά εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά απερίφθη. 52 υπέρ, κατά απερίφθη. 53 υπέρ, κατά απερίφθη. 54 υπέρ, κατά εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά απερίφθη. 56 υπέρ κατά απερίφθη 57 υπέρ κατά απερίφθη 58 υπέρ κα... επαληθεύουμε την 58 δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα Πέντε υπέρ 17 κατά. Σε φέστατα το αποτέλεσμα, αποβιάστηκα. 59 υπέρ κατά Απερίφθη. 60 υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε την 60. 11 υπέρ, 11 κατά. Απερίφθη. 61 υπέρ, κατά. Απερίφθη. 63 υπέρ, κατά. Απερίφθη. 9 υπέρ, κατά απερίφθη 10 υπέρ κατά απερίφθη 11 υπέρ κατά απερίφθη 12 υπέρ κατά απερίφθη συμβαστική 1 υπέρ κατά εγκρίνεται προχωράμε μπροστά Balls 83 υπέρ κατά απερίφθη 84 υπέρ κατά εγκρίνεται. 85 υπέρ κατά απερίφθη. 86 υπέρ κατά απερίφθη. 87 ε, υπέρ κατά απερίφθη. 88 υπέρ κατά απερίφθη. 89 υπέρ κατά εγκρίνεται. 90 υπέρ κατά εγκρίνεται. 91 υπέρ Επαληθεύουμε την 91. 11 υπέρ, 11 κατά περίφθη. 92. Δύο χωριστές έχω εδώ. Συνομένως σωστό είναι. Χωριστά η 92 και 94. Μαζί, μάλιστα. 92-94 λοιπόν, υπέρ, κατά. Ε, πάλι θεύμα. Τέσσερα μαζί ταυτόσιμες από ό,τι λέει. Α, δεν είναι ταυτόσιμες. Καλώς. Άρα ψηφίζουμε πρώτα το 92. Ναι, έτσι ήταν σημειωμένο και χειρόγραφα πάνω στο χαρτί μου. Φαίνεται ότι είναι τη τελευταία στιγμή. Λοιπόν, 92 Πρώτα, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ούτω ή άλλω δεν τα σαφή τα αποτελέσματα. Τι κάνουμε κατευθείαν ηλεκτρονική. 14 κατά. 8 υπέρ την... Απορρίψαμε το 94 παρακαλώ τώρα. Πάλι ηλεκτρονικά. 11 υπέρ, 11 κατά. Απερίφθη. 93 υπέρ. Κατά. Έχει απορριφθεί. 95 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά. Η πλειοψηφία το δέχεται. 97 υπέρ. Κατά. Απερίφθη. 98 υπέρ έχει καλυφθεί, καλώς, καλώς, καλώς έχουν φύγει και 99 έχει καταπέσει, η 100, παρακαλώ, υπέρ, κατά. Απερίφθη. 101, υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 102, υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 103, υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 104, υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 105, υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 106, υπέρ, κατά. Επαληθεύουμε. Την 106. 12 υπέρ. 10 κατά. Εγκρίνεται 107. Κατά 107. Επαλήθευση. Ε, λείπει μία ψήφος. Έντεκα υπέρ, 10 κατά εγκρίνεται, 108 υπέρ κατά. Επαληθεύουμε την 107 παρακαλώ. 10 υπέρ, 12 κατά απερίφθη. 109 υπέρ, κατά απερίφθη. 63 της ΣΥΜΚΟ υπέρ. 63 ΕΜΚΟ υπέρ, κατά απερίφθη. 110 υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε την 110. 17 υπέρ κατά. Απερίφθη και αυτή. 111 υπέρ κατά. Απερίφθη. 113 υπέρ κατά απερίφθη 112 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 118 υπέρ κατά απερίφθη 119 όχι, α, καλύπτεται ε, έχετε δίκιο σε αυτό και ευχαριστώ για την υπενθύμηση και 37 38 τώρα υπέρ, κατά, απερίφθη, 115 υπέρ, κατά, εγκρίνεται 116, καλύπτεται 118, καλύπτεται 119, υπέρ, κατά, απερίφθη, 120 υπέρ, κατά, επαληθεύουμε την 120. 5, υπέρ, δεκα, 7 κατά νομίζω σαφές το αποτέλεσμα. 121 υπέρ κατά Απερίφθη. 122 υπέρ κατά. Επαληθεύουμε την 122. «12 υπέρ 10 κατά εγκρίνεται, 123 καλύπτεται και τώρα πάμε στην 124 υπέρ κατά. Απερίφθη 125 υπέρ, κατά. Απερίφθη 126 υπέρ, κατά. Απερίφθη 127 υπέρ, κατά. Απερίφθη 128 υπέρ, κατά. Απερίφθη 129 υπέρ, κατά. Απερίφθη 130 υπέρ, κατά. Απερίφθη 131 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 132 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται 133 υπέρ κατά. Εγκρίνεται. Δεν είναι σίγουρο να επαληθεύσουμε λοιπόν. Έντεκα υπέρ, 10 κατά, εγκρίνεται. 134 υπέρ, κατά και αυτό το επαληθεύουμε, 134. Απερίφθη συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 3. Συμβαστική υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 140 υπέρ. Κατά. Απερίφθη 141 υπέρ κατά. περίφθη 23 υπέρ κατά. Επαληθεύουμε. 23. Έντεκα υπέρ, 11 κατά απερίφθη. 1 υπέρ. Επαληθεύουμε την υπαριθμό 1. Απερίφθη 11 υπέρ 11 κατά. 24 υπέρ κατά. Εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά. Απερίφθη 2 υπέρ κατά. Απερίφθη 25 υπέρ κατά. Επαληθεύω την 25. 11 υπέρ, 11 κατά, απερίφθη 27 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται 26 υπέρ, κατά. Την έχουμε καλύψει την 26, 28 με συγχωρείτε λέει ο πρόεδρος, υπέρ, κατά. Απερίφθη 29 υπέρ, κατά. Απερίφθη 3 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται 4 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται 30 υπέρ, κατά ε, απερίφθη 31 υπέρ 31 επαληθεύουμε Έντεκα υπέρ, 11 κατά, απερίφθη. Και πάω στην 5, 32 και 33 υπέρ κατά. Ε, απορρίφθηκαν 34 υπέρ κατά. Απερίφθη 35 υπέρ κατά απερίφθη 36 ε, υπέρ κατά εγκρίνεται 5 της εμικό ταυτόσημη 38 υπέρ κατά επαληθεύουμε την 38 12 υπέρ, 10 κατά εγκρίνεται. Ε, η 37 έχει καλυφθεί. 39 τώρα υπέρ, κατά. Επαληθεύουμε την 39. 12 υπέρ, 10 κατά. Εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά εγκρίνεται 40 καλύφθηκε 41 είχε απορριφθεί 42 υπέρ κατά απερίφθη 43 υπέρ κατά εγκρίνεται 44 υπέρ επαληθεύουμε τη 44 παρακαλώ 10 υπέρ, δέκα κατά. Απερίφθη. 45 υπέρ. Επαληθεύουμε. Επτά υπέρ, 5 κατά. Εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά εγκρίνεται. 48 υπέρ. Τι, γιατί όχι τη 48. Λοιπόν, ψηφίσουμε τη 47. Ήταν λάθο σειρά στον κατάλογο. Υπέρ, κατά. Επαληθεύουμε τη 47. 10 υπέρ, 11 κατά, απερίφθη. Και τώρα η 48 υπέρ, κατά. Επαληθεύουμε και τη 48. 10 υπέρ 11 κατά απερίφθη. Ήμκο 15 υπέρ κατά απερίφθη. 49 υπέρ κατά. Επαληθεύουμε. 49. 10 υπέρ 12 κατά απερίφθη και το σύνολο τώρα με ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. 22 υπέρ, χωρίς αποχές και χωρίς αντίθετες ψήφους. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Τώρα έχω την έκθεση της κυρίας Λίχτεμπεργκ για την εφαρμογή της συνθήκης Λισαβόνας. Έχετε να πείτε τίποτα κυρία Λίχτεμπεργκ. Όχι, ε, τροπολογία πρώτη λοιπόν, υπέρ κατά εγκρίνεται, δύο υπέρ κατά επαληθεύω. Την υπαριθμόν δύο τροπολογία. 11 υπέρ, 11 κατά περίφθη, 3 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται το σύνολο της εκθέσεως ηλεκτρονικά. Είκοσι υπέρ, μία ψήφος κατά και μία εποχή. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Μετά έχουμε την έκθεση της κυρίας Γκαλό. Έχετε να πείτε κάτι, όχι, να ψηφίσουμε κατευθείαν, μάλιστα. 8 λοιπόν, υπέρ κατά, α, εγκρίνεται, 9 υπέρ κατά, εγκρίνεται, 10 υπέρ κατά, εγκρίνεται, 53 υπέρ κατά, απερίφθη, 7 υπέρ κατά εγκρίνεται 12 υπέρ κατά εγκρίνεται 13 υπέρ κατά εγκρίνεται 14 υπέρ κατά εγκρίνεται 15 υπέρ κατά εγκρίνεται 16 υπέρ κατά εγκρίνεται 17 υπέρ κατά εγκρίνεται 54 υπέρ κατά Επαληθεύουμε. 54 παλήθευση. 11 κατά 10 υπέρ. 10 ε, κατά. Εγκρίνεται. 15 παρακαλώ. Αληθεύουμε. 10 υπέρ, 11 κατά απερίφθη, 56 υπέρ, κατά εγκρίνεται, 57 υπέρ, κατά απερίφθη, 58 υπέρ, κατά. Επαληθεύουμε την 58. Δέκα υπέρ, δέκα κατά περίφθη, δεκαοχτώ υπέρ, κατά εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά εγκρίνεται 20 υπέρ κατά εγκρίνεται 21 υπέρ κατά εγκρίνεται 22 υπέρ κατά εγκρίνεται 23 υπέρ κατά εγκρίνεται 59 υπέρ κατά επαληθεύμα 59 επαληθεύση 11 υπέρ 10 κατά. Εγκρίνεται. 60 υπέρ κατά. Το επαληθεύουμε και αυτό. Δέκα υπέρ 11 κατά απορρίφθη. 61 υπέρ κατά. Επαληθεύουμε. 61. Απερίφθη. 62 υπέρ. Παληθεύουμε και αυτό. 62. Με 10 ψήφους κατά εγκρίνεται και περνάμε στην 63 υπέρ κατά εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά απερίφθη. 66 υπέρ κατά εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά. Επαληθεύω την 67. 10 υπέρ, 11 κατά περιφυση. 8 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά εγκρίνεται, η 96 καλύπτεται, 27 υπέρ, κατά εγκρίνεται, 70 καλύπτεται, 28 υπέρ, κατά εγκρίνεται. Η 71 έχει καλυφθεί, 72 υπέρ, κατά εγκρίνεται, 29 υπέρ, κατά εγκρίνεται, 30 υπέρ, κατά εγκρίνεται, 31 υπέρ, κατά Επαληθεύουμε την 31. 13 υπέρ, 9 κατά, εγκρίνεται. 32 ε, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά. Επαληθεύουμε την 33. Εγκρίνεται. Καλύτερα το 73 και πάμε στη 34 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 36 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 37 υπέρ. Κατά. 38 εγκρίθηκε 37. Εγκρίνεται και 38. 39 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 40 υπέρ κατά εγκρίνεται 41 υπέρ κατά εγκρίνεται 42 υπέρ κατά εγκρίνεται 43 υπέρ κατά εγκρίνεται 44 υπέρ κατά εγκρίνεται 40, 74 ε, υπέρ κατά εγκρίνεται 75 καλύπτεται 76 υπέρ κατά καλύπτεται ε, ε επαληθεύουμε 10 υπέρ 10 κατά και απερίφθη 1 υπέρ κατά εγκρίνεται 2 υπέρ κατά εγκρίνεται 3 υπέρ κατά εγκρίνεται 5 υπέρ κατά εγκρίνεται 6 υπέρ κατά εγκρίνεται 7 υπέρ κατά εγκρίνεται 45 υπέρ κατά εγκρίνεται 46 υπέρ κατά, εγκρίνεται 47 υπέρ η 47 καλύπτεται, 48 υπέρ κατά. Επαληθεύουμε τη 48. 10 υπέρ, 11 κατά. Απερίφθη 41 υπέρ, κατά. Απερίφθη 50 υπέρ, κατά εγκρίνεται 52 υπέρ κατά εγκρίνεται και σχέδιο γνωμοδότησης στο σύνολό του υπέρ κατά σας παρακαλώ να και με κάτι σοφορία 11 υπέρ 10 κατά εγκρίνεται η γνωμοδότηση και συγχαρητήρια στην εισηγήτρια Τα οργανωμένα ταξίδια τα έχουμε αναβάλει. Την ψηφοφορία. Και έτσι πάμε στη δική μου πρόταση επιστολής. Έχετε το κείμενο υπέρ, κατά. Αποχές ουδής, εγκρίνατε λοιπόν. Και έτσι. Έχω τώρα μια νομική βάση Επιτροπή Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων. Με την κυρία Ρέγνερ έχετε το λόγο. Αν δεν έχετε πρόβλημα, Πρόεδρε, θα ήθελα να το συστήσουμε πολύ σύντομα. Πρόκειται για τι υπηρεσίε αγορά εργασία 149 είναι η δική μου πρόταση, ως μοναδική νομική βάση. Θέλει κανεί άλλο να λάβει το λόγο, να υπερψηφίσει, να καταψηφίσει. Εγκρίνεται λοιπόν και πάμε στο επόμενο θέμα, πάλι για την, για την κυρία Ρέγνερ με τον καπνό. Ναι, και εδώ θα είμαι σύντομη. Είναι πάντα βέβαια θέμα που γεννά πολύ έντονο ενδιαφέρον η οδηγία για τα καπνά. Και πάλι σύντομα λοιπόν, γιατί θα ήθελα να πω πιο πολλά πράγματα. Έχουμε το φαινόμενο την Κυριακή να εμφανίζονται πάρα, πολλές, ε, πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα στη δουλειά, ε, πάρα πολλά email από τη γραμματεία, και προσπαθεί η γραμματεία βεβαίω να κάνει τη δουλειά τη ε, με πάρα πολύ καλό τρόπο. Εγώ θα ήθελα κατά βάση να είχα τι πληροφορίε πολύ νωρίτερα, ήδη από μια εβδομάδα τουλάχιστον για να μπορώ να μελετήσω προσεκτικά. Θέλω να εκφράσω ρητέ ευχαρισίε στην ε, γραμματεία, η οποία δεν διστάζει και το Σαββατοκύριακο ακόμα να δουλεύει για να κάνει τη δουλειά τη εγκαίρω. Έχουμε στην Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων τη γνωμοδότηση και έχουμε εκφράσει Νομική Επιτροπή τη επιφυλάξει μα προ την νομική βάση. Άρα δεν είναι ζήτημα μόνο εσωτερικής αγοράς. Και εδώ θα κάνουμε μια πρώτα συμβαστική για την ψηφοφορία. Να μην στηριστούμε μόνο στο 14 δηλαδή, αλλά συνολικά και με το 148. Και αυτό για να έχουμε μια στάση συνεπή σε σχέση με τα όσα έχουμε διατυπώσει και με τη γνωμοδότησή μας. Καλώς λέει ο Πρόεδρος, άρα με τις δύο αυτές νομικές βάσεις. Ω, με συγχωρείτε, παρακαλώ φως. Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα ήθελα για άλλη μια φορά να εκφράσω επιφυλάξεις ε, και να επικυρώσω τη συμβαστική πρόταση τη συναδέλφου. Θέλω και εγώ δηλαδή να διατυπώσω ως πολιτική ομάδα της επιφυλάξεις μας, αλλά να δηλώσω ότι θα υποστηρίξουμε τη συμβαστική πρόταση της συναδέλφου. Καλώς λοιπόν, συμπληρωματική νομική βάση, υπάρχουν αντιρρήσεις, όχι, εγκρίνεται και ευχαριστώ την εισηγήτρια. Και τώρα, μετά τα καπνά, έχουμε την υγεία των ζώων. Ε, εδώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Λέει η κυρία Ρέγνερ, είναι τόσο διαφιλονικούμενο το θέμα που θα προσπαθήσω να ακολουθήσω αυτή την πρόταση. Υπάρχουν αντιρρήσεις, λέει ο πρόεδρος, όχι. Καλώς, ευχαριστώ. Τελευταία νομική βάση, λοιπόν. Ζήσαμε οκτώνα, το ίδιο ισχύει. Υπάρχουν αντιρρήσεις, όχι. Εγκρίνεται λοιπόν και έτσι τελειώσαμε και τις νομικές βάσεις. Και πάω στο σημείο 10, κυρία Ρέγνερ, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ναι, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχουμε μια πρόταση τη Επιτροπή λοιπόν για τη θέσπιση μιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελία για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής ΕΑ, ζητήματα τα οποία δεν θα κρυθούν με τη συναπόφαση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόνο σύμφωνη γνώμη μπορεί να δώσει. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία ευτυχώ πλέον ε, σβήνει σιγά σιγά, αλλά ακόμα θα εφαρμοστεί σε αυτήν εδώ την περίπτωση. Γνωρίστε τα δεδομένα. Πρόκειται για ένα ζήτημα πολύ ε, ενδιαφέρον. Έχει προξενήσει πολύ ενδιαφέρον και συζητήσει πολλέ, όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στα εθνικά. 14 εθνικά κοινοβούλια έχουν αξιοποιήσει τη μέθοδο τη κίτρινη κάρτα. Κατάσταση λοιπόν είναι η εξή. Είναι αυτή για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών έχει την καθήλυνα αρμοδιότητα, έχει κάνει την γνωμοδότησή της. Για το άρθρο 86 ως νομική βάση πρόβλημα δεν βλέπουμε. Και ως εκ τούτου θα ήθελα να επικεντρωθώ στο περιεχόμενο, στην ουσία δηλαδή τη γνωμοδότηση. Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών έχει την καθήλυνα αρμοδιότητα, όπω είπα. Έχουμε όμω και την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, δυνάμει του άρθρου 50. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι πολύ σημαντικό, εφόσον ε, γνωμοδοτήσει η Επιτροπή μας, να ασχοληθούμε στα θέματα, με τα θέματα στα οποία έχουμε ακριβώς αρμοδιότητα. Γι' αυτό δεν θέλω να επεκτείνω το πεδίο συζητήσεων για την Επιτροπή μας. Θα συζητήσουμε μόνο τα ε, θέματα αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μας. Άρα έχουμε το 13 της ε, προτάσεως της Επιτροπής, το οποίο ε, αφορά τις ε, ποινικές αρμοδιότητες και εδώ γίνεται μια επιλογή μεταξύ δύο ομάδων ποινικών αδικημάτων. Η μία ομάδα προβλέπει αρμοδιότητα ε, με βάση το άρθρο 12 της παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Αγγελίας αυτεπαγγελτός, ενώ το 13 για ορισμένη κατηγορία ποινικών αδικημάτων μπορεί να αιτιολογήσει παρουσία αρμοδιότητα. Η δεύτερη ομάδα δεν ορίζεται όμως από τον κανονισμό. Πρόκειται δηλαδή για τις πτυχές εκείνες τις οποίες τα εθνικά κοινοβούλια αντιδρούν και αιτιολογημένα βεβαίως ε, και έχουν επιφυλάξεις προς την, ως προς την ε, ε, διατύπωση. Γι' αυτό λοιπόν μια από τις προτάσεις που θέλω να κάνω είναι καταρχάς βελτίωση της ε, διατύπωσης. Έχουμε λοιπόν την ε, περίπτωση της απόπειρας ε, παραβίασης των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οικονομικών συμφερόντων, αυτό το λέω για να είμαστε πιο σαφείς. Μετά έχουμε την προϋπόθεση που αφορά το άρθρο 13 για το αδίκημα ώστε να αφορά τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Το διαγράφουμε αυτό γιατί μπορεί να υπάρχει διάπραξη πολλαπλών αδικημάτων και παραβίαση διαφορετικών κανόνων δικαίου. Μια άλλη πτυχή, μια δεύτερη πτυχή που θέλω εγώ να εισαγάγω είναι η αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Στην πρόταση κανονισμού λοιπόν της Επιτροπής ε, αρμοδιότητα έχουν τα εθνικά δικαστήρια. Εμένα με προβληματίζει αυτό. Μπορεί δηλαδή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αφενός αφετέρου ένα εθνικό δικαστήριο να έχουν διαφορετική τοποθέτηση ως προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και αυτό που με απασχολεί είναι ε, εσείς από τις πολιτικές ομάδες τι θα μπορούσατε να προτείνετε. Δεν θέλω δηλαδή να αφήσουμε περιθώριο για βεβαιότητα. Και γι' αυτό θα ήθελα όσο το δυνατόν πιο σαφής τοποθετήσεις και προτάσεις από τα μέλη της Επιτροπής Τρομικών Υποθέσεων. Στο τρίτο σημείο έχουμε τη δομή και το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί το προσωπικό της Όλαφ αλλά λέει ότι θα πρέπει να εμπλακεί και το προσωπικό της Eurojust. Από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης αναφέρεται η ε, χρήση προσωπικού. Εγώ δεν έχω προτίμηση ούτε για την Eurojust ούτε για την Olaf. Δεν έχω μια προτίμηση. Θα ήθελα να δω εσείς τι έχετε να πείτε λοιπόν. Πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει να βρούμε μια καλή και λογική λύση και βεβαίω, θέλω να ακούσω τη γνώμη τη δική σας των μελών της Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων και η τελευταία παρατήρηση η κατάρτιση των Ευρωπαίων εισαγγελέων. Ο φίλος Λουίτζι Μπερλιγκουέρ, όπω ξέρετε, έχει αγωνιστεί πολύ για την υπόθεση αυτή και έχει καταφέρει σε θέματα κατάρτισης, μετεκπαίδευσης, άνα, έχει κάνει πολύ σημαντική δουλειά και χρήσιμη και για τους Ευρωπαίους Εγγελείς. Αυτά, εν ολίγης, οι πτυχές τις οποίες εγώ θεωρώ κάπως προβληματικές. Αυτά. Θα προχωρήσουμε και θα προγραμματίσουμε και για την προσεχή νομική βάση. Είμαι στη θέσή σας να ακούσω τις προτάσεις σας και τις συστάσεις ε, για θέματα που θα μπορούσα να συμπεριλάβω στο κείμενο. Ευχαριστώ Σπερώνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όσον αφορά την πρόταση αυτή, πολλά εθνικά κοινοβούλια έχουν τοποθετηθεί προβάλλοντας αντίρρηση, διότι λένε ότι δεν σέβεται την αρχή της επικουρικότητας η αρμόδια επιτροπή να κρίνει κατά πόσο συνάδει μια πρόταση με την αρχή της επικουρικότητας είναι η νομική επιτροπή και ήθελα να γνωρίζω γιατί αντιθέτως η δική μας επιτροπή δεν γνωμοδότησε επ' αυτής της πτυχής αλλά ετοιμάζει μια γενικόλογη γνωμοδότηση χωρίς να αξιολογεί πριν την πτυχή της επικουρικότητας. Α, νόμιζα ότι αυτό κάναμε. Το βάλαμε στην ημερήσια διάταξη, το συζητήσαμε. Δεν καταλήξαμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα βέβαια. Είναι ένα θέμα το οποίο τακτικά προκύπτει η επικουρικότητα. Το συζητάει ο συγκεκριτής, η συγκεκριτρία. Όχι απαραίτητα με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θα δούμε με την έκθεση της κυρίας Ρέγνερ. Από εκεί θα προκύψει. Άλλες παρατηρήσεις υπάρχουν. Δεν βλέπω τίποτε προς το παρόν. 24 Ιανουαρίου λοιπόν η προθεσμία... Α, ο κύριος Φως. Παρακαλώ. Ναι, ζητώ συγγνώμη πρόεδρε. Σε σχέση με την Eurojust, θα ήθελα να πω δύο λόγια και νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσει ε, εν γέννη ο τρόπος με τον οποίο ε, θα συνδυαστούν οι εργασίες της Eurojust, της Ευρωπαϊκής Αγγελίας των Εθνικών ενδεχομένω Δομών. Ε, κάπως πρέπει να οργανώσουμε αυτές τις δομές, γιατί συσσωρεύονται διάφορα επίπεδα και τελικά δεν μπορούμε να ε, αποφύγουμε τις επικαλύψεις. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να έχουμε μια σαφή αξιολόγηση για την, και συζήτηση για την κατανομή των αρμοδίτητων. Δεύτερον, η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει το εάν θέλουμε να θεσπίσουμε μία ε, ποινική δικαιοδοσία ή εάν θέλουμε να αφήσουμε την κρίση νομικών θεμάτων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Γιατί εκεί θα έχουμε να κάνουμε και με την ε, κρίση των ενδίκων μέσων ε, στο, ή βοηθημάτων ε, στο δικαστήριο, πράγμα το οποίο σημαίνει προθεσμίες για κατάθεση, συζήτηση και το καθεξής. Αυτά λοιπόν νομίζω ότι δεν μπορούμε ακόμα να τα δούμε σαν συνολική εικόνα και γι' αυτό παρακαλώ να έχουμε το περιθώριο να αναλογιστούμε με προσοχή την κατεύθυνση στην οποία θέλουμε να προχωρήσουμε. Μπορεί να μας αρέσει η κατάσταση όπως έχει τώρα, αλλά θα πρέπει να δούμε με προσοχή πώς θα την αναδιαμορφώσουμε. Και να έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα στοιχεία. Και προσωπικό αν είναι, αν είναι από την Όλαφ, αν είναι από την Eurojust. Και όχι μόνο αυτό, μία σαφή δομή. Και νομίζω ότι και εσείς έχετε δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό. Διαφορετικά θα καταλήξουμε σε ένα απίστευτο πλέγμα αρμοδιοτήτων, επικαλύψεων, δομών ε, που η μία θα καλύπτει την άλλη και δεν θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε αυτό. Ναι και η Επιτροπή το λόγο. Πού είσαστε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σχολιάσω την, ε, το εξαιρετικό σχέδιο έκθεσης της εισηγήτριας και σας ευχαριστούμε που θέτετε αυτά τα ορθά σχόλια, αλλά πρέπει να κάνω κάποιες διευκρινήσεις. Όπως ξέρετε, συνεχίζονται οι συζητήσεις του Συμβουλίου για την πρόταση της Κομισιόν και είναι πράγματι πολύπλοκες οι διαπραγματεύσεις. Το άρθρο 13 είναι σίγουρα ένα από τα θέματα που έχουν συζητηθεί και θα συζητηθούν εκτεταμένα και στο Συμβούλιο και η νομική μας υπηρεσία νομίζω ότι πολύ λεπτομερώς έχει εξετάσει το άρθρο 13 και έκανε μία σειρά καλών προτάσεων. Πολλές από αυτές επαναλαμβάνονται στο σημείο 1, στο λατινικό 1, α, β, γ και δ. Βέβαια έχουμε ένα πρόβλημα στον κατάλογο αυτό που είναι το πρώτο σημείο, το α, τα δικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 13, να είναι μόνο εκείνα που προβλέπονται στις νομοθετικές πράξεις της Ένωσης. Αυτό δεν είναι κατανοητό για μας, γιατί προβαίνεται στη σύσταση αυτή. Εδώ μιλάμε για τα συνδεδεμένα εθνικά δικήματα και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τα δικήματα απάτης. Τώρα η απάτη και τα λογιστικά ε, αδικήματα δεν είναι αρμονισμένα από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε υπάρχει σχετική νομική βάση. Έτσι λοιπόν δεν έχει νόημα το κριτήριο στο α. Το επόμενο σημείο στο 1 είναι το τελευταίο, το λατινικό 3, ότι η Ευρωπαϊκή Συγγελία θα πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά τη από των δικημάτων που έχουν διαπραχθεί που το τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Και το άρθρο 71 της πρόταση θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί πρέπει να περιορίσουμε την αρμοδιότητα της εισαγγελίας ε, μόνο ε, αφού έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία αφού έχει συστηθεί η εισαγγελία, θα λάβει μια σειρά υποθέσεων εισαγγελία που συνήθως συνεχίζονται, δηλαδή θα έχουμε πράξεις που θα έχουν διαπραχθεί πριν από το χρόνο της σύστασης και δεν είναι πολύ τεχνητό να διαχωρίσουμε αυτά τα δικήματα σε δύο κατηγορίες, αυτά που είχαν διαπραχθεί πριν από την θέση λειτουργία και αυτά που διαπράχθησαν μετά. Έτσι λοιπόν εγώ θα σας συνέστηνα να σκεφτείτε αυτό το τρίτο σημείο υπό το ένα. Τώρα, σημείο 3. Που έρχεται μετά το σημείο 1. Πραγματικά εδώ λέτε ότι θα πρέπει να υπάρχει μία συνέπεια σε σχέση με την ε, προσφυγή, με την προσφυγή και θα πρέπει να σχετίζεται με τις παραβιάσεις που έχουν να κάνουν ε, με το θέμα της νομιμότητας ε, της ε, έρευνας ε, και νομίζω ότι και τα εθνικά δικαστήρια και όχι τα ευρωπαϊκά δικαστήρια θα πρέπει να δικάσουν το θέμα των ζημιών. Όμως ε, το σύστημα θα πρέπει να είναι αντίστροφο. Θα πρέπει λοιπόν τα εθνικά δικαστήρια να επισέρχονται εδώ και υπάρχει μια εξήγηση γιατί πιστεύουμε ότι τα εθνικά δικαστήρια είναι καλύτερα για να εκδικ να αξιολογούν το θέμα της νομιμότητας, γιατί τελικά αυτές οι υποθέσεις θα καταλήξουν στα εθνικά δικαστήρια να δικαστούν. Και το τελευταίο σημείο στην παράγραφο 4, λυπάστε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σκεφτεί να μεταφέρει ανθρώπινους πόρους από την Όλαφ. Εδώ δεν μιλάμε για ανθρώπινους πόρους, μιλάμε για οικονομικούς πόρους από την Όλαφ. Υπάρχει παρεξήγηση λοιπόν εδώ. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να μεταφερθούν μια σειρά θέσεων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όμως ε, δεν μιλάμε για ανθρώπους που εργάζονται στην Όλαφ, αλλά για πόρους ε, που αντιστοιχούν σε αυτές τις θέσεις ε, και φυσικά εσείς θα συμμετέχετε στην όλη διαδικασία, στη σύσταση της εισαγγελία. Εμείς προτείνουμε εδώ μία δομή που θα καλύπτει διοικητικέ υπηρεσίε, δεν θα έχει ερευνητέ ούτε εισαγγελίε που θα μπορούν ε, να εργαστούν και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί λοιπόν εδώ. Και για το τελευταίο σημείο, συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει κατάρτιση και στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να έχουμε επαρκεί πόρου για την κατάρτιση των εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ε, έτσι ώστε να μπορούν να ερευνούν τα οικονομικά αδικήματα. Ευχαριστώ, Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για τις προτάσεις και τις υποδείξεις, ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις παρατηρήσεις και τις διευκρινήσεις που μας προσφέρει και προσβλέπω σε μια πολύ καλή συνεργασία που θα επιτρέψει να βαθύνουμε σε όλα τα θέματα. Όμως θέλω να διατυπώσω μια θεμελιώδη τοποθέτηση για τον τρόπο εργασίας η εισαγωγή μιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι μια καταπληκτική ιδέα, μια πολύ καλή προσέγγιση, ένα καλό εγχείρημα, προκειμένου και ο πολίτης της Ευρώπης να έχει περισσότερη εμπιστοσύνη στα νομικά, στα ίσενομες τάξεις, ε, αλλά όχι μόνο αυτό, να μπορεί μέσω της Ευρωπαϊκής Αγγελίας να βλέπει κάτι το απτό. Ωστόσο, υπάρχει ένα ωστόσο ε, παίρνουμε πολύ μεγάλη προσοχή και σοβαρότητα τα, τα λόγια του κυρίου Σπερώνη, ότι δηλαδή μένει δουλειά να γίνει και δεν θεωρώ ευφυές επειδή τελειώνει η θητεία λίγο πολύ να κάνουμε βεβαιασμένες προτάσεις, ειδικά σε θέματα τα οποία μπορούν να διαταράξουν την ε, εμπιστοσύνη στις ένωμες τάξεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε όποια πρόταση μας αρέσει χωρίς προσοχή. Πρέπει να κάνουμε πολύ προσεκτική προετοιμασία και μελέτη. Δεν θέλω λοιπόν ε, να εναντιωθώ στις θέσεις σας, θέλουμε επικοδομητικό τρόπο να προχωρήσουμε και μαζί, αλλά κάποια ζητήματα πρέπει να διευκρινιστούν. Ποια είναι η κατάσταση με την επικουρικότητα, Έχουμε μια σαφή τοποθέτηση για την επικουρικότητα, την έχουμε διατυπώσει δημόσια και τώρα ερχόμαστε με αυτή τη γνωμοδότηση. Πολύ θα ήθελα βεβαίω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προχωρήσει με τη γνωμοδότησή του και να την καταθέσει με την υποστήριξη της συντριπτικής πλειονότητας των μελών του ε, στην αρμόδια καθήλων επιτροπή. Νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για προτάσεις, ουσιαστικές προτάσεις, όχι δευτερεύουσα σημασία, και να προσφέρουμε όχι μόνο ή όχι κυρίως την πολιτική επιλογή αλλά την νομική βάση και την νομική εξειδίκευση ε, στην ε, Καθήλυνα Αρμόδια Επιτροπή. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που με στήριξαν και βέβαια όταν μιλάμε για όλα ξέρουμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ε, πόρους και όχι μόνο οικονομικούς είναι ένας δρόμος τον οποίο μπορούμε να, πάρθ να πάρουμε και νομίζω ότι είναι καλό να αποφύγουμε μαζί με τα χλωρά, να και τα, μαζί με τα ξερά, να καίμε και τα χλωρά, διατυπώνοντας υπερβολικές ε, απαιτήσει. Μπορούμε να έχουμε μια πιο στενή συνεργασία στο Συμβούλιο. Ξέρουμε βέβαια, οι διαδικασίες συνήθως τι φέρνουν, πόσες δυσκολίες φέρνουν και γι' αυτό την γνωμοδότησή μου μπορείτε να περιμένετε να τη διαβάσετε χωρίς όμως ιδιαίτερα ενθουσιώδεις ε, εκφράσεις. Θα αναφέρομαι ασφαλώς τις συνθήκες πλαισίου των μέρους και των μελών και τη διαδικασία αυτή της κίτρινης κάρτας. Θα πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουμε αυτή την ε, παρέμβαση των εθνικών δικαστηρίων και θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίηση και τη χαρά μου για τις όποιες τροπολογίες πρόκειται να κατευθούν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ρέγνερ, δεν βλέπω να ζητεί κανείς άλλο το λόγο. 24 Ιανουαρίου για τις ε, τροπολογίες, 12 το μεσημέρι. Πάω στο σημείο 9. Παρουσίαση της ε, αξιολόγησης επιπτώσεων Κυρία Κεμπάλου, να το λόγο. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε που μας δίνετε το λόγο και τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε αυτή την αρχική αυτή αξιολόγηση. Θα κάνω μια εισαγωγή και ο να αναφερθεί εκτενέστερα στο θέμα να, και θα εξηγήσει τα πορίσματά του ίδιος. Να επενθυμίσω ότι η αρχική αξιολόγηση που έκανε η μονάδα αξιολογήσεω συνεπιών για τι επιτροπέ, είναι μια ρουτίνα, είναι μια αυτόματη διαδικασία. Εντοπίζουμε τα ισχυρά σημεία και τις αδυναμίες μιας αξιολογήσεως αντιχτυπού. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι συνάδελφοι ήδη έχουν εκπονήσει για την Επιτροπή μια έκθεση για το κόστος της ελλείψεως της Ευρώπης. Έχουμε συνεργαστεί μαζί τους Θεωρήσαμε όμως παρόλα αυτά ότι θα ήταν χρήσιμο να δούμε την αξιολόγηση συνεπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σαν κάτι συμπληρωματικό, διότι αυτή η αξιολόγηση συνεπειών θα είναι χρήσιμη καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και όχι μόνο στην αρχή. Γι' αυτό λοιπόν προβήκαμε σε αυτή την εξέταση και θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο. Ευχαριστώ Έλκε. Κλάδιο Κολοβάρ το όνομά μου και εγώ συνέταξα την αξιολόγηση αυτή. Σύντομη θα είναι η παρουσίασή μου. Έρχεται, έχετε το έγγραφο. Είναι διαθέσιμο και στην στοσελίδα της ομάδας προβληματισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ισχυρά σημεία και αδυναμίες. Υπάρχουν πολλά ισχυρά σημεία της αξιολογήσεως συνεπιών. Εντοπίζεται το πρόβλημα ε, ξοδεύουμε χρόνο και χρήμα για να αποδείξουμε την ε, ακρίβεια των εγγράφων, ότι είναι ε, αληθινά έγγραφα. Και μπορούμε να δώσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα για τα προβλήματα. Υπάρχουν επιπλοκές, μια, σε ένα γάμο ε, ουγγροβελγικό και για την υποβολή προσφορών πλευρά εταιριών ή προβλήματα εταιριών να εγκατασταθούν στο εξωτερικό. Για ποιον είναι πρόβλημα αυτό είναι πρόβλημα για 12 εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δίδονται διάφορα αριθμητικά στοιχεία, αλλά ακόμα το 15% ο χαμηλότερος αριθμός, το 15% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είναι αρκετά μεγάλος στόχος για το μέτρο. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι κάτι πρέπει να γίνει και όπως είπε το 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρειαζόμαστε απλούστερες, σαφέστερες και πιο προσβάσιμες διαδικασίες. Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ταιριάζουν με αυτά που ζητά το Κοινοβούλιο. Η εξολόγηση συνεπιών είναι ένα εργαλείο, δίδει στοιχεία για την ενίσχυση των πολιτικών. Θέλουμε συλλογικά σαν ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα καλύτερες επιδόσεις και θα αναφερθώ σε κάποια προβλήματα Θέλουμε απλούστευση της αποδοχής κάποιων δημοσίων εγγράφων. Ποια έγγραφα είναι αυτά. Αυτό δεν αναφέρεται εκτενώς στην αξιολόγηση συνεπιών. Η αξιολόγηση λέει απλώς ότι υπάρχουν κάποια έγγραφα συχνά χρησιμοποιούμενα και παραθέτει κατάλογο περίπου κάποιων εγγράφων που αναφέρονται και στο άρθρο 3. Γιατί επελέγησαν κάποια έγγραφα, δεν εξηγείται αυτό. Θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνονται περισσότερα, λιγότερα έγγραφα. Δεν γίνεται λόγος για τον αριθμό των εγγράφων. Υπάρχει και κάποια μεροληψία όσον αφορά τις επιλογές. Στι επιλογές που έχουν επιλεχθεί και στον τρόπο που παρουσιάζονται. Μικροαπλουστεύσεις γίνονται Υπάρχει δυνατότητα να μην υπάρξει δράση και υπάρχει και ακραία επιλογή, δηλαδή εναρμόνιση των πάντων και σε εθνικό επίπεδο υποχρεωτικά. Δεν είναι κάτι ρεαλιστικό αυτό σαν λύση και υπάρχουν κάποιες άλλες λύσεις που συμπεριλαμβάνονται στην προτίμηση και προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπετε ότι υπάρχει κάποια κλίση προς μία πλευρά και στη διατύπωση και στην παρουσίαση. Θα το δείτε στην αξιολόγηση πιο λεπτομέρο αυτός, αυτό. Λοιπόν, λεπτομέρειες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει πολύγλωσσα έντυπα. Δεν δείτε πλήρης απάντηση πώς θα επιτευχθεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ότι τα έγγραφα που αναφέρονται στο παράδειγμα, τα πέντε, είναι και τα πιο σχετικά για την λύση αυτή, γιατί δεν εξηγεί, θα μπορούσε να παρουσιάσει διαφορετικές επιλογές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν το έκανε, ίσως να υπάρχουν κάποιοι λόγοι γι' αυτό, αλλά δεν εξηγούνται. Τα ωφέλη δράσεως είναι περισσότερα από το κόστος. Ε, αυτό είναι σημαντικότατο και το κόστος εκτιμάται. Υπάρχει τάξεις μεγέθους για τις δαπάνες, για τα έξοδα. Βλέπετε τους υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γίνονται κάποιες υποθέσεις και αυτά είναι τα τελικά στοιχεία. Δεν θα επισέθω σε τεχνικές λεπτομέρειες. Βλέπετε ότι το περισσότερο, το μεγαλύτερο κόστος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλεται στη μετάφραση. Αν περί αυτού πρόκειται, θα περίμενα να δω μεγαλύτερη συμμετοχή των μεταφραστών που θα επηρεαστούν από το μέτρο στις συζητήσεις, διαβούλευση μαζί τους. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Το ψάξα, αλλά δεν υπάρχει. Το Συμβούλιο Μελέτης Αντιχτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζητήθηκε να δώσει ε, λεπτομέρειες και στοιχεία κατόπιν αιτήματος μεταφραστών. Δεν δόθηκαν οι λεπτομέρειες και καμιά φορά εκείνοι που θα θέλαμε να απαντήσουν ε, δεν απαντούν. Ε, υπάρχει διεύθυνση τμήμα, διεύθυνση μετάφραση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα μπορούσε να δώσει χρήσιμες πληροφορίες. Προχωρώντας πάμε σε μια εκτίμηση που δίδεται το, το κόστος η δαπάνα για το χρήση του IMI του συστήματος πληροφοριών για την εσωτερική αγορά Βλέπετε το συνολικό στοιχείο, το σύνολο. Είναι περίπου 600.000 ευρώ το κόστος, πιθανότατα αναέτος. Και αυτό είναι αποτέλεσμα κάποιων υποθέσεων που βλέπετε να εμφανίζονται. Υποθέτουμε βασικά, υποθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι τέσσερις δημόσιες αρχές ανταλλάσσουν πληροφορίες, χρειάζονται μισή ώρα η καθεμία για να προβούν στην ανταλλαγή στοιχείων και αφορά 14.000 έγγραφα ε, ε, και νομίζω που θα, θα ήταν αμφίβολου γνησιότητας. Δηλαδή 1% των ειδικών σφραγίδων των αποστήγων που ανταλλάσσονται στην Ευρώπη, της ειδική θεώρησης. Είναι μέσος όρος είναι 22 ευρώ το κόστος αυτής της ειδική σφραγίδας. Περιορισμένο κόστος αλλά επηρεάζεται πολύ από δύο υποθέσεις. Είναι ευαίσθητο. Δηλαδή, ότι η, χρειάζεται πάντα η ανταλλαγή πληροφοριών μισή ώρα ακόμα και στην αρχή που οι δημόσιες αρχές να μην γνωρίζουν την ύπαρξη του IMI καλά, να μην γνωρίζουν καλά το IMI και όχι μόνο 1% είναι αμφιβολά έγγραφα και το, το IMI που παρουσιάζεται σαν αποτελεσματικό εργαλείο θα χρησιμοποιείται μόνο για τις ειδικές φαγίδες θεώρησης της αποστήγη και όχι για άλλα θέματα που ασχολούνται με την ε, έγκριση, την ε, διαπίστωση της αυθεντικότητας του εγγράφου. Αν το στοιχείο αμφιβολιών πάει στο 2 με 3% θα διπλασιαστούν και θα τριπλασιαστούν οι δαπάνες. Αν συγκρίνουμε με τα στοιχεία που δίδονται στο IMI, 14.000 ε, συναλλαγές τέτοιες είναι πολλές. Βλέπετε στο κάτω μέρος τον αριθμό των συναλλαγών ανταλλαγής πληροφοριών το 2011 λίγο πολύ είναι 3.000. Μάθαμε ότι το IMI είναι ευέλικτο εργαλείο, μπορεί να αντιμετωπίσει μεγαλύτερη ζήτηση, αλλά προκύπτει το ερώτημα. Αν ξαφνικά αυξηθούν οι ανταλλαγές πληροφοριών, θα υπάρξει αύξηση κόστους. Ε, σε αυτή την έννοια είναι καλό που το άρθρο 7 εισάγει ευελιξία, όπως βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια. Μία ευελιξία που δεν φαίνεται να καλύπτεται στην αξιολόγηση αντιχτύπου. Δηλαδή η δημόσια αρχή μπορεί να χρησιμοποιήσει το IMI ή να έρθει σε επαφή με την κεντρική αρχή του κράτους μέλους. Απ' τη μια λοιπόν αυτό ίσως να μειώσει το κόστος για το IMI, απ' την άλλη όμως δεν γνωρίζουμε πόσο θα κοστίσει στη δημόσια αρχή που επιλέγει τη δεύτερη εναλλακτική. Αυτά είναι τέσσερα σημεία που σχετίζονται με τη διαφάνεια. Το πρώτο. Το δεύτερο αφορά τη διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους φορείς. Πρέπει να υπάρχει επαφή μαζί τους. Μετά, αν δίνουμε κάποιες εκτιμήσεις, πρέπει να είναι βάσιμες. Και τέλος, η αξιολόγηση συνέπειων θα πρέπει να αντιστοιχεί στην πρόταση. Όπως έλεγα, εν γέννη η αξιολόγηση συνέπειων είναι μια ισχυρή αξιολόγηση και ελπίζω ότι θα σας βοηθήσει να λάβετε αποφάσεις ως Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς το λόγο, εισηγητής πολύ σύντομα. Έχουμε αποφασίσει, η ιδιαίτερη βοήθεια να μας προσφέρει. Γιατί νομίζω ότι η ψηφοφορία προβλέπεται στην Ολομέλεια την ε, μεταπροσεχή εβδομάδα. Επομένω, ε, χωρί να θέλω να υποτιμήσω τη δουλειά που κάνουμε εδώ πέρα, γιατί πάντα καλό είναι να λαμβάνουμε και συμπληρωματικέ πληροφορίε, θα ήθελα ωστόσο να επισημάνω ότι το θέμα αξιολόγηση συνεπειών το έχουμε συζητήσει εντατικότατα πριν από δύο-τρία χρόνια, αν δεν απατάμε με την κυρία Νίμπλη ως συγκήτρια. Και θα ήθελα να επισημάνω, χωρίς βέβαια να έχει άμεσο η συνάφεια με το συγκεκριμένο θέμα, ότι έχουμε πει πως ε, Οι λόγοι πολλές φορές οφείλονται και στο, στη θεσιμότητα των βουλευτών. Η διάθεση λοιπόν των Προέδρων δεν επέτρεψε να προχωρήσει δεδομένων των συνθήκων τώρα. Το λέω με πολύ διπλωματικό τρόπο. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω την αξία τέτοιου είδους ανταλλαγής απόψεων, θέλω να επισημάνω ότι καλή αξιολόγηση είναι ποιόν, αλλά την απόφαση, επειδή είναι και πολιτική, την παίρνουμε εμείς. Έτσι προβάλλω στην εξή παρατήρηση. Στο άρθρο 3 αναφερθήκατε στην αρχή της τοποθέτησής σας. Είναι και η αιτιολόγηση της Επιτροπής, η οποία προβαίνει σε μια αξιολόγηση συνεπιών. Λέει ότι δεν υπάρχει αξιολόγηση και μας εξηγεί με αυτό το επιχείρημα την επιλογή της να καταθέσει τα έγγραφα με αυτόν τον τρόπο. Πολιτική απόφαση όμως και εγώ συγητής ε, δεν το κοίταξα περισσότερο. Ξεκίνησα από τα, πραγματικότητα. Η πραγματικότητα τι μας λέει, ότι ο πολίτης έχει κάθε δικαίωμα, γι' αυτό άλλωστε είμαστε και εμείς εδώ, να δει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει όταν πάει να αισθήσει ένα έγγραφο σε ένα άλλο κράτος μέλος να αντιμετωπίζονται. Και μάλιστα η απόφαση, όπως είπαμε, είναι πολιτική. Προτείνω λοιπόν. Δεν κατάλαβα πρόκειται για μια πρώτη προσέγγιση. Προτείνω λοιπόν να το επεξεργαστούμε περαιτέρω. Τρίτη φορά νομίζω θα το πω σήμερα. Να το πάμε στο προσεχές κοινοβούλιο, στην προσεχή θητεία γιατί θα ολοκληρωθεί η πρώτη ανάγνωση χωρίς κινητικότητα από πλευρά του Συμβουλίου και πρέπει να πω ότι έχω λάβει και από πλευρά του Συμβουλίου παράκληση ούτε καν να ψηφίσουμε, να ψηφίσουμε ούτε καν εδώ ούτε στην ε, Ολομέλεια, γιατί φαίνεται κάποια κράτη-μέλη έχουν κατατρομάξει από αυτήν την ε, κατάσταση, ότι δηλαδή είναι σοβαρή η προσέγγιση μας. Μπορεί να μην γελάμε, αλλά είναι έχουν τρομάξει από αυτή τη σοβαρή προσέγγιση και θα βόλευε πολύ το Συμβούλιο να ανταθεί στο θέμα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να τον θαρρύνουμε μαζί με την Επιτροπή, πέραν των λεπτομεριών, να προχωρήσει με, το δεύτερο, με την επόμενη θητεία μετά τις εκλογές σε μια δεύτερη ανάγνωση. Και έτσι μπορούμε να έχουμε τις πληροφορίες για να προχωρήσουμε σε μια ουσιαστική αξιολόγηση. Το να κατατρομάξει κανείς το Συμβούλιο ήδη καλό το βρίσκω. Σπερώνει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την έκθεση αυτή και θα ήθελα να προσπαθήσουμε να πάμε πέρα από την προσέγγιση που παρουσιάστηκε. Πράγματι υπάρχει μια δυσκολία στο να αναγνωρίσουν διάφορα κράτη ένα πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σε μια άλλη χώρα. Έτσι λοιπόν πρέπει να προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε τη ζωή των πολιτών ακόμη και αν ένα από τα προβλήματα που έχω ακούσει είναι ότι όταν μια χώρα ζητά ένα πιστοποιητικό και ένας πολίτης, ε, όχι της ίδιας χώρας, δεν μπορεί, ε, το χάρη, να βρει αυτό το πιστοποιητικό γιατί δεν υπάρχει ένα τέτοιο πιστοποιητικό στη χώρα του. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει, το χάρη, στο Βέλγιο ένα πιστοποιητικό που λέγεται ΜΕΡ και δεν υπάρχει στην Ιταλία αντίστοιχο αυτό το πιστοποιητικό. Έτσι λοιπόν, όταν η Ιταλία ζητά το λεγόμενο πιστοποιητικό κατά της μαφίας, στις άλλες χώρες δεν υπάρχει. Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε και αυτή την πτυχή. Όμως ίσως θα έπρεπε να πάμε και πιο πέρα, όπως είπα στην αρχή, γιατί θεωρώ ότι στην Ιταλία έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ στο θέμα αυτό. Από το 2012 στην Ιταλία η δημόσια δίκηση δεν ε, ζητά πλέον πιστοποιητικά από τους πολίτες. Ε, βέβαια, τα πιστοποιητικά ε, λένε στην Ιταλία ότι το παρόν πιστοποιητικό δεν μπορεί να δοθεί προωθεί σε οργανισμούς δημόσιας ε, δηλαδή η ίδια δημόσια διοίκηση πρέπει μέσω του δικού, των δικών της μέσων να ε, μπορέσει να επαληθεύσει τα στοιχεία που υπάρχουν. Ε, εγώ λοιπόν αν δηλώσω ότι έχω γεννηθεί τότε, ότι μένω στην τάδε διεύθυνση και ότι έχω γεννηθεί στην ε, τάδε πόλη, δεν πρέπει να παρουσιάσω και ένα πιστοποιητικό, γιατί η αρχή η οποία ενδιαφέρεται να γνωρίζει αυτά τα δεδομένα, αν είναι αληθή, είναι η αρμόδια η οποία μέσω του συστήματος που διαθέτει η δημόσια διοίκηση ελέγχει αν όσα έχουν δηλωθεί ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματική οδός ε, να κάνουμε τη ζωή πιο εύκολη στους πολίτες. Ε, όχι τώρα να παράγουμε διάφορα πιστοποιητικά που θα αναγνωριστούν λοιπά. Η δημόσια διοίκηση, ακόμη και της αλλοδαπής, είναι αυτή που θα έπρεπε να αναλάβει. Έτσι λοιπόν θα μπορέσουμε να κάνουμε κατανοητό ότι δεν είναι γραφειοκρατική η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν, ε, αν θέλει να μάθει κάτι, η βελγική κυβέρνηση σε σχέση με μένα να πρέπει να μπορεί να στραφεί στις ιταλικές αρχές χωρίς να χρειαστεί εγώ να υποβάλω διάφορα έγγραφα. Έτσι, θα διευκολύναμε τη ζωή των πολιτών ε, και πραγματικά θα τους κάναμε λιγότερο εχθρικούς απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως δυστυχώς εδώ δεν αντιμετωπίζουμε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ακριβώς αυτό είναι και το πρόβλημα ε, που αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά. Ωστόσο θα ήθελα λίγο να αναφερθώ στην εκτίμηση αντικτύπου. Καλό βέβαια όταν έχουμε τέτοιου είδου ζητήματα ή τόσο να προβαίνουμε σε μια πικριτική προσέγγιση της ε, εκτίμησης αντικτύπου από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι και στο θέμα του κόστους βλέπουμε να εμφανίζονται κάποιες παράδοξες εκτιμήσεις. Και μου έχει συμβεί να λέω τέτοιου είδους αλγόριθμο με τα μαθηματικά που έχω κάνει εγώ τουλάχιστον δεν έχω ξαναδεί. Δεν μου φαίνεται κάπως παράξενο όλα αυτά. Ε, το ένα είναι αυτό λοιπόν. Το δεύτερο, σε σχέση με το κόστος. Πολύ ωραία η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, απασχολείται να αξιολογήσει το τι κόστος μπορεί να συνεπιφέρει μία ε, επιλογή ή άλλη. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι το μόνο επιχείρημα. Ιδάλλως πολλά πράγματα θα μπορούσαμε και να τα καταργήσουμε τον, ε, από το κοινό πεδίο τον κοινό χώρο. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορεί να είναι κύριο επιχείρημα ή μοναδικό επιχείρημα το κόστος για πολλά ζητήματα. Ε, λάθος επίσης μου φαίνεται, δηλαδή όταν έχουμε να κάνουμε τα νομικά ζητήματα, να τα προβάλλουμε με τόση επιμονή και μένει το εξής ερώτημα πλέον. Έχουμε μία δυνατότητα μόνο για εκτίμηση αντικτύπου Ερωτώ λοιπόν ποιος επιλέγει για ποιο θέμα θα προχωρήσει η αξιολόγηση αντικτύπου. Δεν είναι σαφής και διαφανής για μένα αυτή η κατάσταση. Εάν λοιπόν είναι κάτι τόσο αυθαίρετο, τότε παίρνει κανείς τον πειρασμό να σκεφτεί ότι η εκτίμηση αντικτύπου μπορεί να επιλέγεται με κριτήρια πολιτικά για να από σαρθρωθούν ορισμένες επιλογές πολιτικές ή ακόμη και να ε, ζημιωθεί πολιτικά ένας ε, επίτροπος. Λοιπόν, θα μου πείτε με ποιο τρόπο γίνεται αυτή η επιλογή, έχουν οριστεί κάποιοι κανόνες, κάποιες συνθήκες με βάση τις οποίες γίνεται αυτή η εκτίμηση. Γιατί τότε είναι πολύ καλά. Αλλά το να μην υπάρχει τίποτα και μετά απλώ να προχωρούμε στην εκτίμηση αντικτύπου και να προβαίνουμε σε μια ανάληψη επαφών με τον ε, ενδιαφερόμενο, τότε μου φαίνεται ότι δεν κάνουμε τίποτα. Δεν ήθελα λοιπόν μια ε, πληροφόρηση. Για το θέμα το ίδιο, βεβαίως και είναι περίπλοκο θέμα. Το έχουμε δει και σε διαφορετικά, διαφορετικούς τομείς ε, και ένομες τάξεις, Φερρυπίν με την Ιταλική, ένομη τάξη με ένα ε, ένομο σύστημα κρατών της Βόρειας Ευρώπης που είναι κάπως αυτόνομα σχέση με το ευρωπαϊκό. Έχουμε δει αυτή τη δυσκολία ότι δεν είναι δυνατόν δηλαδή να εξετάσουμε όλες τις παραμέτρους. Και έτσι πολλές φορές λέμε «Α, επειδή το, η τάδε ένωμη τάξη δεν επιτρέπει να παρέμβουμε, καλύτερα να μην κάνουμε τίποτα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα». Άρα θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να κάνουμε την αλλαγή ή όχι. Εάν μου πείτε ότι τρομάζει το Συμβούλιο με μια νέα πρόταση, θα απαντήσω ότι και εμένα με κατατρομάζουν ε, οι αντιευρωπαϊκές τοποθετήσεις που εκφράζονται με τόση ε, αυτοπεποίθηση από πλευράς του Συμβουλίου. Δεν μπορεί αυτό να είναι μια τοποθέτηση νομική και, εν πάση περιπτώσει, δεν βλέπω κανένα είδου κριτήριο σε σχέση με την εκτίμηση. Ο κύριος Ράπκα χωρί μικρόφωνο. Ναι, και επιπλέον, σε εμά εκπρόσωποι των ομοσπόνδων κρατηδίων μπορεί να έχουν μια τραυματική εμπειρία επειδή ε, κάποιοι άλλοι συνάδελφοί τους από ένα άλλο ομοσπονδοκρατήριο έχουν παρεμποδίσει την λήψη μιας πολύ σοβαρής και σωστής απόφασης. Τέτοιου είδους τραυματικές εμπειρίες έχουμε και στις ομοσπονδιακές χώρες. Εν πάση περιπτώσει, ε, πρέπει να ξέρουμε με ποιο τρόπο λαμβάνονται αποφάσει για ποιο θέμα, με ποιους όρους για την εκτίμηση αντικτύπου. Και αν δεν είναι σωστή ή δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία, τότε πρέπει να βρούμε μια διαδικασία. Ο Πρόεδρος, πριν προχωρήσει στους επόμενους ομιλητές, λέει ο Πρόεδρος, ε, υπάρχουν πολύ σαφείς ε, κανόνες. Η διάσκεψη των Προέδρων ε, σαν ένα εποπτικό συμβούλιο επαληθεύει. Υπάρχει ένα εγχειρίδιο 90 ημέρες μετά αυτά, όλα είναι η έκθεση Νίμπλερ και θα σου στείλω το αντίγραφο αν θέλεις. Ε, γίνεται η κατάρτιση του καταλόγου, η γραμματεία πάει στην αρμόδια επιτροπή, λαμβάνονται οι αποφάσεις με βάση τις προτάσεις των εισηγητών, του εισηγητή ή της εισηγήτριας. Οι συντονιστές ρυθμίζουν κρεμότητες και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτή είναι η κατάσταση. Και τώρα έχω την κυρία Τάιν, την κυρία Νίμπλερ και συνεχίζουμε. Κυρία Τάιν. Ναι, γιατί πρέπει να είναι πολύ γλώσσο το ένα ή το άλλο φυλάδιο ή έντυπο, νομίζω δεν χρειάζεται να το μελετήσουμε, είναι σχετικά αυτονόητο να λέγαμε τη χρησιμότητα. Ε, συμφωνώ με τον κύριο Ραπκάη. Το άλλο που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν υπάρχουν ε, ε, παραπομπές στην νομοθεσία. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε στην περίπτωση, χωρίς να κινδυνεύει κανείς να πτωχεύσει, στην περίπτωση των μικρών εκείνων εντύπων που μπορεί να διαχειρίζεται ένα, μια μικρή υπηρεσία με ένα δεχομένο γραφείο, έναν υπάλληλο ή δύο το πολύ, όπως γνωρίζουμε εμείς και στη Γερμανία, ιδιαίτερα στο Βερολίνο, και που μπορούν να έχουν ε, ίσως όχι μεγάλες ενώσεις συμφερόντων και εκπροσώπους, πρέπει να μπορούν να προχωρήσουν χωρίς να φοβούνται ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με την ανεργία. Εκείνοι που έχουν μεγαλύτερα γραφεία και μπορούν να εργαστούν σε περισσότερες γλώσσες μπορούν να μεταφράζουν και τα πιο ε, μακροσκελή έγγραφα. Τα μεγαλύτερα γραφεία λοιπόν μπορούν να πάρουν τα μεγαλύτερα έγγραφα από 100 σελίδες και πάνω Η έρευνα αυτή έχει μια διάσταση οποία, η οποία με απασχολεί ιδιαίτερα. Είναι η παραποίηση του εγγράφου ε, και δεν τοποθετούμε για τη σφραγίδα της Χάγης, ε, γιατί είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως καλύπτουν πολλές ε, διακρατικές συμφωνίες και σε σφραγίδα της Χάγης πολύ σπάνια χρειάζεται να καταλήξουμε. Αλλά, αλλά όλη αυτή η επαλήθευση ότι δεν υπάρχει παραποίηση εγγράφου, γιατί έχω μιλήσει με εκπροσώπους των αρχών της πατρίδας μου, ξέρω το λέω ότι ισχύει για τη Γερμανία τουλάχιστον, ότι μπορεί να εκδώσουν ένα έγγραφο χωρίς να ε, του περάσει ποτέ από το μυαλό ότι μπορεί αυτό τελικά να φτάσει σε κάποιο άλλο ευρωπαϊκό κράτος να χρησιμοποιηθεί. Ακόμη και από το, δικαστή, από το Υπουργείο Δικαιοσύνη μπορεί να εκδοθεί ένα έγγραφο χωρίς να ξέρουν ότι θα προχωρήσει έτσι. Γι' αυτό λοιπόν και μπορεί να προκύψουν πολλά παραποιημένα έγγραφα και να προχωρήσουν σε άλλες αρχές κράτους μέλους. Γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω πώς μπορούμε να κάνουμε μία ε, να διατυπώσουμε μια επιφύλαξη όπου βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα ή ότι υπάρχουν, εμφανίζονται μαζικές παραποίησεις χωρίς να θέλω βέβαια να ε, κατονομάσω κανένα κράτος μέλος και να γίνω δυσάρεστη, υπάρχουν κράτη στα οποία εμφανίζονται μαζικά παραποίηση εγγράφων. Και απασχολούν αυτά μετά τις αρχές, τώρα έχουμε φτάσει στο ληξιαρχείο της ε, πατρίδας μου, ε, που έχει να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους καταστάσεις ε, σχετικές με υπηκόους άλλου κράτους που μένουν και έχουν ε, παντρευτεί εκεί και θα ήθελα να μου πείτε τι δυνατότητες υπάρχουν να επαληθεύσει μία αρχή, ένα λεξιαρχείο, την γνησιότητα ενός εγγράφου τρίτου, άλλου κράτους, Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο του κατατίθεται. Επίσης από τη μελέτη ε, θα ήθελα να επισημάνω, γιατί και ο συμβολεογράφος το έχω δει πολλές φορές, ε, ότι δεν δίνονται αρκετά λεπτομερείς παρατηρήσεις για τα στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνει η ληξιαρχική πράξη γέννηση ή θανάτου. Δεν έχω καμιά επιφύλαξη ως προς το αν η εκδούσα αρχή, αρχή είναι η βουλγαρική, το βουλγαρικό ή το ρουμανικό ή το ληξιαρχείο κάποιες άλλες ε, χώρας, αλλά πρέπει να υπάρχουν αρκετά στοιχεία νομίζω για να ε, μπορούμε να προχωρήσουν. Δεν καταλαβαίνω γιατί τα κρατη θέλουν να συνεργαστούν. Για τον κύριο Σπερώνη και την ε, περίπτωση που αναφέρει, πολύ καλή ιδέα και νομίζω εύχριστη εξυπηρετεί τον, ε, τον πολίτη γιατί θα πρέπει εκείνος να τρέχει για να βρει τα στοιχεία, τα, τις ληξιαρχικές πράξεις και το καθεξής όταν στη διάθεση του κράτους του υπάρχουν όλα αυτά. αλλά πρέπει να πω ότι στη Γερμανία δεν θα ισχύει αυτό που ισχύει στην Ιταλία. Έχουμε καταρχάς πολλούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν, παντρεύτηκαν, χώρισαν, πήραν διζύγιο. Έχουν ενδεχομένω εγκατασταθεί μαζί με κάποιον σύντροφο σε ελεύθερη σχέση, έχουν ε, ξεκινήσει άλλη οικογένεια και για τους οποίους δεν υπάρχουν στοιχεία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ή και πριν ακόμη έχουμε τις περιοχές σε που από τη ε, Γερμανία πέρασαν στη Γαλλία και μετά ε, έχουν έρθει οι άνθρωποι στη Γερμανία. Έχουμε ζητήματα ε, πράξεων που έχουν τελεστεί από ιερέα και άρα θα πρέπει να καταφεύγουμε στα σχετικά έγγραφα της Εκκλησίας. Έχουμε πολύ αυστηρά όρια μεταξύ των ομόσπονδων κρατηδίων και δεν υπάρχει κεντρικό μητρό στη Γερμανία σε βαθμό που μπορεί κανείς ε, να πει ότι ένα, ε, ε, ένα παιδί μπορεί να μην βρίσκει που έχουν τελέσει το γάμο τους ίδιου του οι είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές να αναστήσει κανείς στοιχεία, έγγραφα, πληροφορίες, ακόμα και για τη δική του την οικογένεια, λόγω της ομοσπονδιακής δονημής. Και γι' αυτό είναι μια υπόθεση η οποία θα κρατήσει πολύ για να προχωρήσει όπως θέλουμε. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει και βέβαια όσον αφορά το αστικό δίκαιο αλλά και στα εμπορικά ζητήματα να υπάρχει μία κάλυψη τουλάχιστον για αυτούς οι οποίοι έχουν μικρότερα γραφεία όπου υπάρχει δυνατότητα για μεγαλύτερες υπηρεσίες μπορούμε να πούμε ότι ζητούμε ε, τις μεταφράσεις κτλ. Αλλά ασφαρώς ε, δεν χρειάζεται πάντα να είναι όλα με αυτούς τους όρους μεταφρασμένους. Κυρία Λίμπλερ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις επί τη βάση των συζητήσεων που προκύπτουν, που είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Καταρχάς ευχαριστώ την ομάδα, τη μονάδα μάλλον εκτίμηση αντικτύπου. Και πάνω απ' όλα για την αντιπαραβολή με το κείμενο της Επιτροπής. Είναι χρήσιμο αυτό. Επίσης, πολύ ενδιαφέρον το ανέφερε και ο κύριος Ραπκάη, μας εξήγησε ποια είναι η διαδικασία στο Συμβούλιο, ότι έχει παρακολουθεί η εξέλιξη και ότι θα χρειαστεί να φτάσει μέχρι το προσεχές Κοινοβούλιο η υπόθεση αυτή. Νομίζω όμως ότι είναι χρήσιμο να μην εγκαταλείψουμε αυτή την προσπάθεια. και να δούμε από τη μία αρχή στην άλλη εάν μπορεί να γίνει η αποστολή, η αίτηση και η ζήτηση εγγράφων από τη μία ε, ε, υπηρεσία στην άλλη απευθείας, από το ένα κράτος μόλις στο άλλο, χωρίς παρεμβαστού πολίτη, ώστε να είναι και γνήσια τα έγγραφα και βέβαια στα όσα είπε η κυρία Τάιν έρχεται το ζήτημα των παραποίησεων που είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το αναπτύξει περαιτέρω η μελέτη αντικτύπου. και να δούμε βεβαίως εσωτερικά ή εξωτερικά τι χρειάζεται περαιτέρω να γίνει. Τι σημαίνει όμως η παραποίηση για την ασφάλεια των αγράφων. Υπάρχει ή δεν υπάρχει, μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αυτό πρέπει να το συμπληρώσετε στην ε, έκθεση. Όπως είπαμε, ίσως δεν θα τα καταφέρουμε σε αυτή την ε, θητεία να το καλύψουμε το θέμα. Αλλά οι δύο που ανέφερα είναι πολύ σημαντικές και θα πρέπει να τη συμπεριλάβουμε σε πραγματεύσεις μεταξύ Βουλίου και Κοινοβουλίου. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, κύριε Ραπκάη. Ε, δεν, ήθελα, δεν είχα μέχρι τώρα την ευκαιρία να προσφέρω τίποτα περισσότερο στη συζήτηση. Κύριε Σπερώνη. Ευχαριστώ. Ζήτησα το λόγο κατόπιν ε, της αναφοράς της συναδέλφου στο κόστος της μετάφρασης. να καταλαβαίνω τις ανησυχίες αυτές. Ε, μπορούμε να πούμε ότι κάποιος κερδίσει και κάποιος χάνει. Δηλαδή, αν κάποιος πρέπει να πληρώσει ένα μεταφραστή, κάποιος ε, κερδίζει χρήματα, αλλά κάποιος πρέπει και να πληρώσει το μεταφραστή. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ε, ως έναν βαθμό ότι μόνο για να διατηρούμε κάποιες θέσεις εργασίας ε, θα πρέπει να βάλουμε τους πολίτες να πληρώνουν ε, κάτι που δεν χρειάζεται. Θα σας πω ότι στην Ιταλία δεν Έχουμε επίσημο επάγγελμα μεταφραστή, οποιοδήποτε μπορεί να μεταφράσει και αν η δημοσιορχή απαιτεί τη μετάφραση ενός εγγράφου, αφού λέγεται σε υποσημείωση ότι είναι πιστή η μετάφραση του πρωτοτύπου και υπάρχουν και ποινικέ κυρώσεις, ακόμη και κράτηση αν κάποιος προβεί σε ψευδείς δηλώσεις. Έπρεπε εγώ πρέπει χάρη να παρουσιάσω ένα βελγικό έγγραφο στην Ιταλία, ένα πρόβλημα δεν υπήρχε, το μετέφρασα εγώ ίδιος και έγραψα ως υποσημείωση ότι ήταν πιστή μετάφραση του πρωτοτύπου, δεν υπήρχε πρόβλημα. Και αν ε, είχε μεταφραστεί με τρόπο μη πιστό, τότε μπορεί να υπήρχαν ε, ποινικέ κυρώσει. Και στην Ιταλία αυτό το σύστημα χρησιμοποιούμε για το αυθεντικό των εγγράφων. Δηλαδή, αν ε, ένα ε, άνθρωπο εγγυάται ότι είναι αυθεντικό το έγγραφο, κατόπιν αν προβεί σε πλουστοποίηση του εγγράφου, τότε όπω γνωρίζετε υπάρχει αδίκημα και υπάρχει και τιμωρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ σύντομα σε σχέση με τη διαδικασία που ακολουθήσαμε στο έργο μας. Υπάρχει κάποια σύγχυση νομίζω σε σχέση με το τι κάναμε εδώ. Κάναμε μια αρχική αξιολόγηση της ε, μελέτης αντικτύπου της Κομισιόν. Δηλαδή ένα πολύ σύντομο έγγραφο που γίνεται στην αρχή της διαδικασίας συνήθως. Όμως ε, εδώ λόγω ε, διάφορων αιτιών έγινε λίγο αργότερα. Όμως αυτό το κάνουμε συστηματικά για κάθε μελέτη αντικτύπου. Δηλαδή το τελευταίο έτος έχουμε παράξει 70-80 τέτοια έγγραφα και έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα. Συνήθως δεν παρουσιάζουμε τα έγγραφα αυτά σε συνεδριάσεις των Επιτροπών, αλλά στην περίπτωση αυτή μας ζητήθηκε να το κάνουμε. Όμως ε, συνήθως ε, δεν πάμε παραπέρα από το να γίνει ένα γρήγορο έλεγχο τη μελέτη αντικτύπου για να σα δώσουμε μια αρχική ιδέα των ισχυρών και των αδύναμων σημείων. Φυσικά, εμείς περιοριζόμαστε στη μεθοδολογία της μελέτης αντικτύπου. Επομένως, δεν λαμβάνουμε τις αποφάσεις αντί για σας. Απλώς παρουσιάζουμε κάποια στοιχεία για τη συζήτηση όλα όσα υπερβαίνουν αυτό, δηλαδή περαιτέρω αξιολογήση τη μελέτη αντικτύπου ή σε σχέση με ένα συμπληρωματικό έργο με μία τροποποίηση που συμπληρώνει τη μελέτη αντικτύπου τη Κομισιόν γίνεται αυστηρά βάση απόφαση των συντονιστών τη αρμόδιας επιτροπή. Εμεί δεν το κάνουμε αυτό ποτέ με δική μα πρωτοβουλία. Και το εγχειρίδιο λέει ότι πρέπει να υπάρχει ευρεία πολιτική συνένεση. Επομένως, οτιδήποτε υπερβαίνει αυτές τις αρχικέ αξιολογήσει πρέπει να βασίζεται σε απόφαση της αρμόδιας επιτροπής. Ευχαριστώ. Καλώς, ευχαριστώ. Έτσι ολοκληρώσαμε τα θέματα μας για σήμερα. Κύριε Τάιν, θέλετε κάτι ακόμα. Πολύ στόμα θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Σπερώνη ότι δεν πρόκειται για παραποίηση ε, στην μετάφραση, γιατί και αυτό είναι βέβαια ποινικό, αλλά στην, ε, στο ίδιο το έγγραφο. Και μπορεί δηλαδή να παραποιηθεί το έγγραφο ως προς την υπογραφή του υπαλλήλου ή τη σφραγίδα, της Υπηρεσία κτλ. Και δεν αναφερόμουν στη μετάφραση. Καλώς λέει ο Πρόεδρος, τώρα κλείνει η συνεδρίαση. Τρεις Ξεκινάμε με κεκλεισμένο των θερών συνεδρίαση και μετά έχουμε και τον Έλληνα Υπουργό.